Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας αρχίσουμε αμέσως. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτησή μας με την ανταλλαγή απόψεων, το διαρθρωμένο διάλογο. Και αυτή τη φορά έχουμε την Επίτροπο κυρία Ελισμπιέτα Μπιανκόφσκα, Επίτροπο Ιστορικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντικά τμήματα αυτά, κρίσιμα θα έλεγα του δικού μας κατοφυλακίου από πολλές απόψεις και πρώτη φορά έρχεται η Επίτροπος φέτος στην Επιτροπή μας. Για φέτος ρε πρώτη φορά. Ναι, αλλά με μεγάλη έκπληξη το διαπιστώνω. Ιούνιο φτάσαμε για να έρθετε πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Ε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα θέματα μας ε, συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα δικά σας, κυρία Επίτροπε, και έχουμε ε, βέβαια ε, να κάνουμε με την απασχόληση, με τις θέσεις εργασίας, με την ανταγωνιστικότητα κτλ. Η δική μας Επιτροπή κάθε φορά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μαθαίνει για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τομείς ευαίσθητους όπως είναι η χαλιβουργία, στρατηγική για τις μικρομεσαίες κτλ. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Our space policy. Galileo, Copernicus. Και βεβαίω το διάστημα, Γαλιλαίος, Κοπέρνικος λοιπά. Επίσης η Ήτρε ενδιαφέρεται ε, πάρα πολύ παγίως για τα θέματα αυτά. Αρκεί να σας αναφέρουμε τις δύο πρόσφατες προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα, ήταν η μία, και η δεύτερη για το σιδηρόδρομο και τα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Την περασμένη Πέμπτη στο Στασβούργο συζητήθηκαν. Ε, δηλαδή ήδη πριν από πέντε μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δίνει συνέχεια οπωσδήποτε σε αυτά τα σημαντικά θέματα και στις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε εμεί πολλά πράγματα, ούτε να μακρηγορήσουμε. Ε, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να συνεχίσει και στα δύο θέματα ιδιαίτερα ε, για την βιομηχανία που παρέχει σιδηροδρομικό υλικό οι προμηθευτές πριν από πέντε μέρες επαναλαμβάνω το εγκρίναμε, τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη και η διαστημική πολιτική της διαστημικής βιομηχανίας εξίσου σημαντική. Και πάλι καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ, για να σας ακούσουμε μεγάλη προσοχή. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα στα πλαίσια του τρίτου διαρθρωμένου διαλόγου με την Επιτροπή σας. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η ημερομηνία αυτή αποφασίστηκε από την Επιτροπή και όχι από μένα. Αυτά ως ε, απολογία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία μας συνάντηση, διότι πραγματικά τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου που σας αφορούν είναι πάρα πολλά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολλά από αυτά. Καταρχάς θα επικεντρωθώ στη βιομηχανία και τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να παίξει μεγάλο ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Καταρχάς όμως θα ήθελα να είμαι σαφής για το εξής. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν γίνεται λόγος για βιομηχανία, δεν εννοούμε μόνο τις ε, επιχειρήσεις και τις κατασκευαστικές. Όπως είπε ο Πρόεδρος, αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις νέες ε, υπηρεσίες, δίκτυα, βιομηχανικές πλατφόρμες, ανάπτυξη ικανοτήτων με τα ποιητική βιομηχανία και επίσης για τις νέες υπηρεσίες προς τους ε, χρήστες, για μηχανήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το σύστημα στο σύνολό του, στη συνολική του αξία και να δούμε και το συνολικό αποτέλεσμα αυτού του συστήματος. Χρειάζεται επίσης μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση από το να εξαρτόμαστε από μεμονωμένα νούμερα. Χρειάζεται... παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε. Ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν. Και αυτό πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας. Θα γνωρίζετε ίσως τα αποτελέσματα από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, από το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες, από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο ρόλος μου λοιπόν τον πρώτο χρόνο της θητείας μου ήταν να συγκεντρώσω όλα αυτά τα ε, έγγραφα στρατηγικής και αυτό και έκανα. Πρόσφατα εγκρίθηκε μια ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Αυτό που θέλουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη σε επενδύσεις, σε εξυγχρονισμό και σε ανανέωση της βιομηχανίας μας. Στις 19 Απριλίου εγκρίθηκε αυτή η ανακοίνωση ως ε, ένα μέρος της δράσης μας για να διευκολύνουμε τους ε, παράγοντες της βιομηχανίας για να ψηφιοποιηθούν. Το, υπάρχει ένα σύστημα τυποποίησης ε, το οποίο χρειάζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας δημοσιεύσαμε ένα σχέδιο τυποποίησης για τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας ως μέρος μιας προσέγγισης που εστιάζει σε πέντε τομείς. 5G, ε, κυβερνοασφάλεια, ε, ασφάλεια των δεδομένων και η τυποποίηση των τεχνολογιών ICT δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο. Χθες συναντήθηκα με πάρα πολλού ενδιαφερόμενους φορείς και συζητήσαμε μια κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση στον τομέα αυτό. Μπορώ να πω ότι η βιομηχανία καλωσόρισε αυτή την πρωτοβουλία για τυποποίηση όλων των συστημάτων, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα πολύ γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Δεύτερο στοιχείο είναι προώθηση συνεργασίας ανάμεσα στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, με τη δημιουργία πλατφόρμας ψηφιοποίησης που θα βοηθήσει και θα δώσει όθηση στις επενδύσεις. Επίσης, χρειάζεται να εξετάσουμε το δυναμικό των μεγάλων δεδομένων, διότι υπάρχει ακόμα αρκετή ε, ασάφεια δικαίου και χρειάζεται λοιπόν να εξεταστούν όλες οι πτυχέ του. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, σε διάστημα βιομηχανία και διάστημα, η διαστημική πολιτική της Ένωση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό ε, μαζικών δεδομένων στον χώρο του διαστήματος. Τα προγράμματά μας, όπως το πρόγραμμα Κοπέρνικος, ε, δημιουργούν τέτοια δεδομένα. Μας ε, δίνει πολλές πληροφορίες για ε, διάφορα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην χρήση της γης και θα δώσει και στην Ευρώπη το δικό της σύστημα πλοήγησης. Οι επιχειρήσεις θα, έχουν, θα αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα δημιουργώντας, δημιουργώντας έτσι νέες υπηρεσίες. Τις επόμενες δεκαετίες θα δούμε μεγάλη πρόοδο στους τομείς αυτούς. Και τον περασμένο μήνα είχαμε την εκτόξευση δύο ακόμα δορυφόρων του συστήματος Γαλιλαίος και στα τέλη περίπου του χρόνου θα είμαστε στη θέση να πούμε ότι μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα Γαλιλαίος. Φυσικά πρέπει να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να επενδύσουν στο διάστημα και να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες. Όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, αυτή τη στιγμή Επεξεργαζόμαστε τη νέα διαστημική στρατηγική σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και θα μας βοηθήσει αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα για το διάστημα στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου. Η στρατηγική αυτή ακόμα βρίσκεται υπό επεξεργασία και αναμένεται να εγκριθεί τον Οκτώβριο φέτος. Εκτιμώ ότι θα καλύψει ε, τους εξής τομείς Καταρχάς, μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικος, ανταπόκριση στις ανάγκε, Τρίτον, που είναι πολύ σημαντικό για μένα ως Επίτροπο, ε, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, τόνωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Διαστήματος, εστίαση στις ε, στρατηγικές πτυχές και επίσης τέλος τη διεθνή διάσταση. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να πούμε ότι θα έχουν ωφέλη τα οποία θα γίνουν αισθητά μόνο όταν ε, συμμετέχουν όλοι και ο δημόσιος τομέας και οι ιδιώτες χρήστες. Χρειάζεται φυσικά να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, το οποίο προβλέπεται για φέτος το φθινόπωρο, σκοπός του οποίου είναι να δημιουργηθεί μία βάση στη βιομηχανία. Μία βάση η οποία θα μπορέσει να απαντήσει στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε κατακαιρματισμένη προσέγγιση στην Ευρώπη. Και αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στηρίζει και θα προσπαθήσει να βρει τρόπους να στηρίξει έργα τα οποία θα δώσουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές φυσικά πολιτικές και σε συνεργασία με, την με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Επίσης, να πω ότι για τον προϋπολογισμό του 2017 θα προτείνουμε προπαρασκευαστικές δράσεις στο χώρο της άμυνας και εάν η πρόταση αυτή στεφθεί με επιτυχία, ενδεχομένως να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη προγραμμάτων ερευνητικών προγραμμάτων για την άμυνα. Φυσικά για να στηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία θα χρειαστούμε τα σωστά εργαλεία, έτσι ώστε να είμαστε αξιόπιστοι και να στηρίξουμε την άμυνα στην Ευρώπη. Η έρευνα είναι το πρώτο στάδιο αυτού του σχεδίου. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σίγουρη πως μπορώ να στηριχθώ σε εσά για τη στήριξή σας. Τώρα. Επόμενος κλάδος που ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός είναι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση κτλ. Για τον λόγο αυτό θα συσταθεί μια ειδική ομάδα υψηλού επίπεδου με ορίζοντα το 2020, διότι χρειαζόμαστε όραμα και σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς και μαζί του και η αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα και να προσπαθήσουμε μέσω της ε, ομάδας αυτής να συγκεντρώσουμε όλους τους ε, αρμόδιους φορείς και γι' αυτό αυτό το θέμα αφορά τα χαρτοφυλάκια πέντε επιτρόπων του Επιτρόπου Έτινγκερ, της Επιτρόπου Μπούλτς και άλλων τριών επιτρόπων. Τώρα, φυσικά το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρήπων δείχνει τα όρια του συστήματός μας με την μη συμμόρφωση των προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αντιδράσουμε γρήγορα και να φροντίσουμε έτσι ώστε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση για τον νέο κανονισμό σχετικά με την έγκριση οχημάτων θα βοηθήσει να βελτιωθεί η ανεξαρτησία των ε, φορέων ελέγχου και η βελτίωση του μηχανισμού για ανακλήσεις οχημάτων και κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να φροντίσουμε όλοι να τηρούν τους νόμους. Ελπίζουμε και εσείς να εγκρίνετε την πρόταση γρήγορα, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας, όπως θα πω και στο Συμβούλιο. Χρειάζεται να δράσουμε γρήγορα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της ε, βιομηχανίας. Και εδώ θα σταθώ στην παγκόσμια υπερχωρητικότητα και στο καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πολύ σαφέ ότι η Κίνα δεν αποτελεί η οικονομία τη αγορά. Γι' αυτό χρειάζεται να βρούμε λύσει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Εργαζόμαστε πήρα το πάνω σε αυτό. Αλλά θα σας πω μόνο ότι στις 21 Ιουλίου θα συζητηθεί το θέμα στο Σώμα των Επιτρόπων και θα υποβάλω προτάσεις. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο, αυτό θα είναι φυσικά το επιθυμητό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε ε, πώς θα προχωρήσουμε και να αναπτύξουμε τα δικά μας ε, αμυντικά μέσα. Χρειάζεται να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που διαθέτουμε, καταπολεμώντας τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τώρα, σε σχέση με την υπερχωρητικότητα προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ε, βασικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις έχω βοηθήσει στη σύσταση μιας συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επίπεδου. Θα συνεδριάσει την επόμενη Δευτέρα, θα συζητηθεί η ενεργειακή πολιτική, οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, το καθεστώς οικονομίας της αγοράς ε, της Κίνας και οι κρατικές ενισχύσεις στον κλάδο. Επίσης, ε, καλωσορίζω την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, της ε, Επιτροπής σας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ καλή η προσπάθεια που κάνετε να σταματήσει αυτή η προσέγγιση κατά αυτή η προσέγγιση σιλό όπως λέμε. Και εμείς από μεριά μας προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανανεώσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες και τις δυνατότητες συνεργασίας. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά τα θέματα. Προσπάθησα να αναφερθώ σε ελάχιστα από αυτά, στα κυριότερα, δεδομένου του λίγου χρόνου που έχω, και να σας ενημερώσω για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Πρέπει βέβαια να πω ότι εστιάζουμε σε ένα ευρύτατο φάσμα και στις μεγάλες και στις μικρές επιχειρήσεις και σίγουρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποφεληθούν περισσότερο από τις πρωτοβουλίες μας. Ε, και να σας πω επί τη ευκαιρία ότι φέτος το φθινόπωρο θα ε, δημοσιεύσουμε μία πρόταση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα, βιομηχανική πολιτική. Είναι το τελευταίο στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών μας. Αν θυμάστε, έστειλα μια επιστολή στα κρατημέλη. Φέτος είχαμε την ανακοίνωση για την έξυπνη βιομηχανία, την οποία θα ακολουθήσει το πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση. Καθαρή βιομηχανία, φέτος το φθινόπωρο. Θα είναι μέρος του ε, πακέτου για την κυκλική οικονομία και του χρόνου. Νομίζω πως μετά από όλα αυτά θα είμαστε πανέτοιμοι για να ολοκληρώσουμε την ε, περιεκτική μας στρατηγική. Θα ενώσουμε όλα τα κομμάτια του παζλ και θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στην πολιτική μας. Θα δούμε πώς μπορούμε τα επόμενα χρόνια να βελτιωθούμε. Ίσως να πω και κάτι ακόμα. Δύο λόγια λοιπόν σε σχέση με αυτά που συνέβησαν δύο μέρες πριν ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, στο Ορλάντο. Πρώτα απ' όλα, όπως ε, και χθες και προχθές το έκανα, ε, θα ήθελα πραγματικά να αποτίσω φόρο τιμή ε, στα θύματα και να εκφράσω στι οικογένειε και τους συγγενεί τους τα συλληπιτήρια. Ε, ξέρω ότι δεν ασχολείται η τούτη εδώ η Επιτροπή με τα πυροβόλα όπλα βάσει της προτάσεω της Κομισιόν έτσι όπω αυτή υπευλήθη έξι μήνες πριν. Ωστόσο πραγματικά θυμίζω ότι εμεί από πλευρά Κομισιόν είχαμε προτείνει την πλήρη απαγόρευση διάθεση της αγοράς των ημιαυτόματων ε, όπλων. Το συζητούμε αυτό λοιπόν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο ε, βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές ε, επιφυλάξεις. Αλλά εδώ μιλάμε για την ε, ασφάλεια των πολιτών και τέτοιου είδους ημιαυτόματα όπλα δεν έχουν θέση στα χέρια των απλών πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος Μπούζεκ και επομένως ε, τώρα να ξεκινήσουμε ε, με τους συντονιστές ε, από πλευράς των πολιτικών ομάδων, κύριος Κάριντς από πλευράς του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θα κάνω πρώτα μια γενική φύσεως ερώτηση. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε και όλα αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία αλλά ξέρετε ότι έχουμε μια ε, στρατηγική ε, ε, σχετικά με τον στόχο του 20% για την επαναβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί και δικό σας στόχο. Επομένως, γενική ερώτηση. Τι κάνουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τον στόχο αυτό. Τον πλησιάζουμε, τον προσεγγίζουμε, είμαστε ακόμα μακριά. Ποια είναι τα αποτελέσματα, πού βρίσκεται η δημιουργία διαθέσεων απασχόλησης και πόσες από αυτές θα αφορούν την παραδοσιακή βιομηχανία γιατί και η βιομηχανία αυτή καθεαυτή αλλάζει ε, διαρκώς και ε, ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξουν κάποιοι ε, ορισμοί. Επομένως, η ερώτησή μου εν είναι τι συνέβη με αυτόν τον στόχο του 20% της επαναβιομηχάνησης, δηλαδή κατά 20% της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Δανίκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, ένα πρώτο σχόλιο. Χαίρομαι που σας βλέπω ε, στην Επιτροπή μας καταρχάς και σας καλωσορίζω. Και δεύτερο, θα ήθελα να εκφράσω κάποια δυσφορία και δυσαρέσκεια ε, γιατί δεν είχαμε εκπροσώπους της DG Growth στη συζήτηση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Όλες οι συζητήσεις ήταν ενδιαφέρουσες, όλα τα ενεργειακά ζητήματα συζητήθηκαν διεξοδικά, αλλά προφανώς ε, ε, έχουν τις πληροφορίε κάποιοι άλλοι και όχι εμείς πάντα. Ε, έγινε μια μελέτη σκοπιμότητας ε, για την ενέργεια και μιλάει για πιθανή αύξηση κατά 20% των τιμών της ενέργειας. Μα δεν είχαμε συμφωνήσει να μειωθεί. Πώς μιλάμε για αυξήσεις τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι ο πληθυσμός και η βιομηχανία και η βιοτεχνία θα πρέπει να προσανατολίζονται στο 20% γιατί 60% ε, των ε, Ευρωπαίων έχει υπολογιστεί ότι ζουν πλέον σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Αυτά τα έχετε λάβει υπόψη σας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη ε, του άνθρακα. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το τι θέλετε να κάνετε για το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ε, υπάρχει δυνατότητα ο άνθρακας να είναι καθαρός. Τα τελευταία τρία χρόνια ε, η Γερμανία, ας πούμε, έχει επιλέξει να προχωρήσει προς μια πράσινη οικονομία του άνθρακα. Στη Ρουμανία τι θα γίνει με τα ανθρακοριχεία, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες, όπου το επόμενο διάστημα, την επόμενη τριετία, θα χάσουν τη δουλειά τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αν αυξηθεί και κατά ένα ευρώ η τιμή των πιστοποιητικών, για ε, το δηλαδή για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, θα αυξηθεί κατά ένα ευρώ η κιλοβατόρα. Σας έχω στείλει επανειλημμένα επιστολές για τη χαλιβουργία. Μιλάτε για νέα ορόσημα και benchmarks, πολύ ωραία. Μα εδώ πρόκειται για το 10% ε, των ε, εργοστασίων. Πού βρίσκονται αυτά, μπορείτε να μας τα πείτε. Ποια είναι αυτά τα εργοστάσια που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές και για την ανταγωνιστικότητα αυτή τη μετράμε σε κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ελπίζω η συνάδελφος Γκρίφιν τώρα να μην θυμώσει αν πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να συνεισφέρει σε συγκεκριμένες αποζημιώσεις ε, που θα πρέπει να καταβάλλονται ε, σε κάποια ε, εργοστάσια στη Ρουμανία. Δηλαδή τώρα θα φέρουμε τις χώρες αντιμέτωπες, θα κλείνουν τα εργοστάσια στη μία χώρα και θα σώνονται σε άλλη. Για το ETS επαναλαμβάνω, θέλαμε να είχε υπάρξει διαβούλευση πολύ ε, πιο έντονη. Είπατε ότι χρειάστηκε να συναντήσετε πάρα πολλούς. Κανένα ευρωβουλευτή θέλετε να συναντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι σου που έχω την ευκαιρία να ε, συζητήσω με την ε, Επίτροπο. Θα ήθελα να πω στην κυρία Μπιανκόφσκα κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται πολύ ε, σοβαρά. Πρώτα απ' όλα τα χαλιβουργία. Η χαλιβουργία λοιπόν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είπατε κι εσείς ότι το πρόβλημα είναι ότι η Κίνα δεν είναι χώρα με οικονομία αγοράς. Ερώτηση λοιπόν στο μέλλον. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Κατανοώ ότι σε κάποια άλλη συνεδρίαση ίσως μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι δύσκολο και περίπλοκο. Ε, ε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο χαλιβουργικός κλάδος είναι εξαιρετικά ε, μεγάλες και τις έχουμε αναφέρει συχνά εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτό όσον αφορά το χάλιβα. Έχω και κάτι άλλο, ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιό σας είναι ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος. Αυτά τα δύο προγράμματα λοιπόν. Ερώτηση, ερώτηση. Πώς θα σταθεροποιηθεί ε, η σχετική υπηρεσία, όπως είπατε και εσείς, σχεδόν ε, το ίμιση των δορυφόρων ε, θα ε, φτάσουν σε μια πολύ δύσκολη φάση και μάλιστα θα εκτοξευτούν τέσσερις τον Σεπτέμβριο. Πιστεύετε ότι είναι πιθανόν, είναι δυνατόν να προωθήσετε ε, ακόμα περισσότερο ε, κυρίως ε, τον Γαλιλαίο έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία. Επίσης αναφερθήκατε σε ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός αυτό του Ορλάντο και αναφερθήκατε στην νόμιμη κατοχή ημιαυτομάτων όπλων. Αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα. Εγώ κατανοώ ότι εδώ ε, ε, υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι. Απ' την άλλη πλευρά, η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή περιλαμβάνει πολλές ασάφειες ε, και ελλείψεις ισορροπιών που στο μέλλον μπορεί να καταλήξουν σε πολύ δυστάρεστες καταστάσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα σε νομοθετικό ε, επίπεδο. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε τώρα περισσότερα προβλήματα. Ε, ε, νομίζω ότι αντί να ξεκινάμε από την αρχή δημιουργώντας ενδυνάμει προβλήματα, καλύτερα θα ήταν να αντιγράψουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες ε, ας πούμε ε, για την κατοχή όπλων, πυροβόλων ε, ή μη αυτομάτων για την αποθήκευση κλπ. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν βασιζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Κύριε Σιλικιώτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπα, ε, αρχικά πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Βεβαίω τίθενται πολλοί στόχοι. Ε, δεν ακούσαμε πολλά πράγματα όμως για την σημερινή κατάσταση στη βιομηχανία και της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια κατάσταση που είναι σε κρίση κυρίως κατά την άποψη λόγω των πολιτικών της σκληρής λιτότητας. Λόγω των πολλών ετών κρίσης και ύφεση, η διαδικασία αποβιομηχανοποίηση ιδιαίτερα του Νότου εντείνεται, ενώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει κλείνουν μια μετά την άλλη. Όσε δεν καταφέρουν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να προβούν σε καμιά επένδυση, ενώ συνεχώς προχωρούν αναγκαστικά σε απολύσει, σε μειώσει προσωπικού. Ε, έτσι, κατά νέα όψη μα, ακυρώνεται οποιαδήποτε προοπτική για ανάκαμψη και ανάπτυξη προ κοινωνίας. κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, γι' αυτό και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Όσον διάφορα το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο παρουσιάζεται ω απάντηση σε όλα τα προβλήματα, δυστυχώ δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ιδιαίτερα στι χώρε που βρίσκονται σε παρατεταμένη νυχεσή, όσο στηρίζεται στι ιδιωτικέ επενδύσει που έχει σαν στόχο να μειώσει το ρίσκο του. Η ομάδα μα, η ΓΚΟΕ, είναι ξεκάθαρο πω αυτό που χρειάζεται για μα είναι να αυξηθούν οι δημόσιε επενδύσει με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα κράτη-μέλη, να ενισχυθεί η πολιτική των κρατικών επιδοτήσεων. Έτσι θα στηριχτεί ουσιαστικά η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μέχρι σήμερα ε, δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά, κονδύλια, ακόμα και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, στήριξη, για στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, και ελάχιστα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, κυρίως της βιομηχανίας. Κυρία Επίτροπε, είναι καλή η ψηφιοποίηση, το μέλλον, η προοπτική, η αξιοποίηση του διαστήματος, η έξυπνη βιομηχανία. Το ζητούμενο είναι θα έχουμε σε κάποιες περιοχές της Ένωσης βιομηχανία για να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις νέες ε, Γιατί η εικόνα που βλέπουμε σε πολλέ περιοχέ τη Ένωση είναι ότι υπάρχει μια πλήρη αποβιομηχανοποίηση και διαλύονται βιομηχανίε, κυρίω οι μικρομεσαίε. Εξίσου σημαντικό κατά την άποψή μα είναι να υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που όπω όλοι γνωρίζουμε είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα ανάπτυξη, να ληφθούν υπόψη οι ανάγκε του στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και να προωθηθούν μέτρα για διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Κυρία Επίτροπε, αναφερθήκετε στο σκάνδαλο με τους ρήπου, αλλά το ζήτημα πάντα είναι να δρούμε προληπτικά και όχι εκ των υστέρων. Δηλαδή έπρεπε αυτό το σκάνδαλο να προληφθεί και όχι να προσπαθούμε εκ των υστέρων να διαμορφώσουμε και να, ε, νέους κανόνες. Ε, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα, ε, Προ την κατεύθυνση τη στήριξη πραγματική οικονομία τη βιομηχανία, θα ήθελαμε να ακούσουμε αν υπάρχουν ε, πιο συγκεκριμένα μέτρα από την Κομισιόν. Επίση, ποιε ρυθμίσει θα προσθέσετε για να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME. Έχουμε ξανακούσει σε αυτή την Επιτροπή ότι θα πάρετε κάποια μέτρα για, ε, για ενίσχυση αυτού του προγράμματο. Και τέλο, θα θέλαμε να ακούσουμε πιο συγκεκριμένα ποια μέτρα θα προωθηθούν για να υπάρξει στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπίσουν τον αθέμητο ανταγωνισμό που θα επιφέρει η Διατλαντική Επενδυτική Εμπορική Συμφωνία, η Συμφωνία TTIP. Είναι γνωστό ότι αυτή η συμφωνία ενδεχομένω να πλήξει κύρια τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχουν κάποιε σκέψει για να αντιμετωπιστούν όλε αυτέ οι αρνητικέ επιπτώσει που θα επιφέρει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν τοποθετήσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων από τους συντονιστέ και πάμε στους υπολείπους ομιλητέ, Ο κύριος Πίπερ, ο πρώτος ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε περιμένουν εναγωνίωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο TTIP και δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω να επιταχύνετε όσο μπορείτε να προχωρήσετε γιατί ε, αυτό θα είναι όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω τρία σχόλια. Πρώτον, η κατάσταση ανταγωνισμού σε σχέση με την Κίνα. Εκεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουμε τεράστια προβλήματα. Είτε πρόκειται για παραγωγής κεραμικής ή για προμηθευτές ε, στον τομέα του αλουμινίου ή του χάλιβα, οι μικρές εταιρείε δεν τολμάνε. Σου λένε εκεί υπάρχει dumping και μπορούν να το αποδείξουν, αλλά οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ μακροχρόνιες και δεν τολμάνε να το καταγγέλουν οι εταιρείε. Αν ε, συνεχιστεί αυτό τώρα για μήνες, φοβάμαι ότι σε πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη, λόγω αυτή της ανίποτης και ανήκουστης κατάστασης ανταγωνισμού από την Κίνα θα μπουν λουκέτα σε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρακαλώ επιταχύνετε τις διαδικασίες του ανταγωνισμού. Δεύτερη ε, παρατήρηση, ενεργειακή απόδοση. Την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσουμε εάν θα έχουμε στόχο εξοικονόμησης όχι ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση της τάξης του 40%. 40% είναι το μισό της ε, κατανάλωσης ενέργειας σχεδόν. Εκεί ε, εγώ υποστηρίζω τη θέση, όπως και πολλοί άλλοι, ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πληγούν. Παράδειγμα, Θέλουμε να περάσουμε στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, να έτσι να κυκλοφορούμε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκεί θα χρειαστούμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας, τελική ενέργεια και θέλουμε να τις ε, αποθηκεύουμε από τις ανανεώσιμες. Και τώρα έρχεστε και λέτε 40% εξοικονόμηση. Έτσι παρεμποδίζουμε την πρόοδο, την καινοτομία και τις θέσεις εργασίας. Και θα παρακαλούσα μια δήλωση της Αρμόδιας Επιτρόπου για τη Βιομηχανία. Τελευταία παρατηρήση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μάλιστα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται. Εχθές ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας μάλλον, και μας λένε ότι, εντάξει, είναι επιπλέον ε, κίνητρο της Εθνικής ε, Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπάρχουν έργα στη Γερμανία, στην Πολωνία και αλλού και projects που θα πρέπει εμείς να τα ε, προβάλλουμε και να τα διαφημίζουμε. Στη Γερμανία δεν ξέρει ψυχή ε, τι είναι το ΕΦΣΙ. Εμείς εδώ τσακωνόμαστε για το ΕΦΣΙ και ε, σπάζω κεφαλιάζουμε, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν άγνοια απόλυτη για το τι εστί ΕΦΣΙ. Καλό θα ήταν λοιπόν να προβάλλουμε και να διαφημίζουμε και τα καλά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ και για τις πολλές δραστηριότητε. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω μόνο σε ένα σημείο. Η προώθηση και ενίσχυση της βιομηχανίας είναι κάτι που ενδιαφέρει πολλούς συναδέλφους. Αυτό δεν γίνεται μόνο με ίδια μέτρα. Μπορεί να σημάνει και ελαφρύνσεις ή μάλλον και προφύλαξη από την υπερβολική ρύθμιση, να μην φορτώνουμε πάρα πολύ τη βάρκα και να μην εμποδίζουμε τη δουλειά τους. Μιλήσατε για τη χαλιβουργία, ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Στη χαλιβουργία έχουμε το θέμα της Κίνας, έχουμε και θέματα εμπορικά, αλλά έχουμε και το εξή γεγονός. Με το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχουμε δημιουργήσει τόσο κακές προϋποθέσεις, ώστε ο Χάλιβα στην Ευρώπη σχεδόν δεν έχει καμία τύχη καμία πιθανότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει καμία ευκαιρία, γιατί εσείς είστε μία επίτροπος και μόνο. Μπορείτε να πείσετε και άλλους συναδέλφους. Να είναι πιο ευνοϊκή η ρύθμιση για τη βιομηχανία. λύσει υπάρχουν και θα μπορούσαν να βρεθούν. Παράδειγμα. Να, ε, δεν λέω να πειράξουμε το στόχο για το κλίμα και να ενισχύσουμε Αλλά ε, τα πιστοποιητικά και τις άδειες τώρα τα έχουν δει τα κράτη ως πλουτοπαραγωγική πηγή για να ε, γεμίζουν τους ε, κρατικούς κορβανάδες. Ξέρω ότι το Συμβούλιο αφίσταται, αλλά θα μπορούσε το Συμβούλιο να καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συζητούν, κάνουν πρόταση, βγάζουν κάποια σημεία και έχουμε ένα περιθώριο ελιγμό και χειρισμών για τη βιομηχανία. Αυτό θα βοηθούσε τη χαλιβουργία πολύ περισσότερο από όλα αυτά τα ωραία λόγια και τα μεγαλόστομα που ακούμε εδώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Και εγώ ερώτηση για την Κίνα έχω. Η Κίνα πραγματικά έχει εξαιρετικά επιθετική στάση. Ακούμε ότι ε, ε υπάρχει ένα θέμα με το, την εταιρεία Κούκα που κατασκευάζει ρομπότ και πρόκειται να εξαγοράσει τη Γερμανία. Δεν θέλουμε ε, εμείς να πούμε κάτι διαφορετικό, αλλά πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την επεκτατική στρατηγική της Κίνας. Δεν θα πρέπει να τονίσουμε την αμοιβαιότητα. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε κύριε Επίτροπε. Ξέρω ότι θα συζητήσετε με τους συναδέλφους. Έχετε άποψη πριν πάτε σε αυτή τη συνεδρία, σε δική σα θα με ενδιαφέρε. Και πολύ συγκεκριμένα μια ερώτηση για το σιδηρόδρομο. Ε, σε μια ερώτηση του Κοινοβουλίου που κάναμε την περασμένη Πέμπτη και τη συζητήσαμε στην Ολομέλεια, δεν απαντήσατε τίποτα γιατί απουσιάζατε. Και κατά τα άλλα αυτό το επικρίνω εγώ ως φόδρα. Όχι για την προσωπική σας απουσία, αλλά γιατί δεν ήταν κανένας επίτροπος που να έχει την παραμικρή σχέση, έστω και κατά διάνοια, με το σιδηρόδρομο. Που είναι για αυτή η επίτροπη και δεν ήταν κανείς από αυτούς παρών. Άρα ε, το θεωρώ αυτό μεγάλη ασέβεια προς το Κοινοβούλιο. Και σας ερωτώ πότε πρόκειται να έχετε ένα διάλογο ε, με τη βιομηχανία ε, που παράγει υλικό για το σιδηρόδρομο, γιατί και αυτά 400.000 θέσει εργασία είναι και εργαζόμενοι. Μην μιλάμε μόνο για τη Χαλιβουργία. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε ειδική ε, συνεδρίαση για εκείνους που παράγουν υλικό για το σιδηρόδρομο. Τι θέλετε να κάνετε εκεί και τι συνέχεια θα δώσετε στο ψήφισμα που εγκρίναμε την περασμένη Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόερ, Τόγια. Ευχαριστώ. Ε, γεια σας κυρία Επίτροπε. Κοιτάξτε, μια συλλογική καθολική στρατηγική για τη βιομηχανία είναι πάρα πολύ επίγουσα. Εσείς είπατε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, θα φέρετε του χρόνου μια τέτοια ε, στρατηγική. Αλλά ε, υπάρχει ένα συλλογικό πλαίσιο, αλλά δεν θα πρέπει να το περιμένουμε. Υπάρχουν και τρέχουσες καταστάσεις. Πρώτον, ε, τι γίνεται με το ε, ορίζοντα. Υπάρχουν ε, πολλές βεβαίως αιτήσει. Τι γίνεται με το ΕΦΣΙ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι γίνεται με την έρευνα και την και τεχνολογική καινοτομία. Δηλαδή είναι η έρευνα που μεταφράζεται σε προϊόν που φτάνει στην κατανάλωση. Ας πούμε, γίνεται με τις κοινοπρασίες στην ηλεκτρονική. ε, καλή καινοτομία, καλή έρευνα, αλλά πώς θα βοηθήσουμε τα προϊόντα να φτάνουν στην αγορά. Οπότε σας ερωτώ το εξής και σε σχέση με αυτή τη στρατηγική που θα μας φέρετε για τη βιομηχανία, εν αναμονή αυτής, πώς μπορούμε να συντονίσουμε κάπως τη χρήση των διαφόρων μέσων και εργαλείων που έχουμε, που θα πρέπει από τώρα να χρησιμοποιούνται, γιατί είναι κατεπήγον το θέμα της ε, ε, βιομηχανίας και πώς θα επαναβιομηχανίσουμε ε, την Ευρώπη. Ας πούμε, η κυρία Βέρνερ μιλούσε για τον σιδηρόδρομο. Υπάρχουν τομείς που είναι ηγετική δύναμη Ευρώπη, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί έχουμε λίγο κατακαιρματίσει τις προσπαθίες μας και χάνουμε ε, δυνάμεις, πάει ο κόπος χαμένος, δεν θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε, να συντονίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Μας ε, εξαγγέλλεται σήμερα ένα πλαίσιο και μια στρατηγική, αλλά από σήμερα μπορούμε να κάνουμε τίποτα στην Ευρώπη για να ξεπεράσουμε τον γκάπ, αυτό το χάσμα που μας χωρίζει από άλλες ε, περιοχές του κόσμου και να μην μείνουμε πίσω. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκανε. Βεβαίω θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Είναι στόχος μας αυτός που έχει να κάνει με το ΑΕΠ, 20% του ΑΕΠ να παράγεται από τη βιομηχανία και αυτό σημαίνει αποφασιστική δράση όμως από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να βρούμε νέες ευκαιρίες, νέες αγορές, όλα αυτά που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπο σήμερα. Ιδιαίτερα η πολιτισμική βιομηχανία που παρόλες τις οικονομικές ε, δυσκολίες που έχουμε δημιουργεί θέσεις εργασίας. Και εδώ γίνεται λόγος και για τα δικαιώματα, τα πνευματικά, τα συγγενικά, γιατί εάν δεν έχουμε πραγματική πολιτιστική βιομηχανία που να πληρώνεται και να υποστηρίζονται η παραγωγή και η δημιουργή σωστά, τότε θα χαθεί ή θα αποδυναμωθεί. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα δεδομένα. Ε, τα αναφέρατε ως ευκαιρία. Εντάξει, μπορεί να είναι ευκαιρία αυτό, η ε, εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων, αλλά υπάρχει και το θέμα της ιδιωτικής ζωής και σφαίρας και πώς αυτή θα προστατεύεται. Ε, αναφερθήκατε σε ένα θέμα και εσείς και κάποιοι συναδελφοί που είναι η απειλή ε, της χαλιβουργίας. Εμείς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αλλά θα πρέπει να αναλάβετε δράση απέναντι στην Κίνα και στον τομέα του χάλιβα. Επίσης, είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύει τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αυτό αφορά και τις εταιρείες που είναι πολύ ενεργοβόρες, όπως μπορεί να είναι η βιομηχανία αλουμινίου, χάλιβα κτλ. Για το ETS εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό κοινωνικό ταμείο που να αποζημιώνει αυτούς τους κλάδους λόγω του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Αλλιώς έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό στο εσωτερικό το ίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς διότι υπάρχουν κράτη που έχουν ιδίους πόρους και μπορούν να ε, βοηθούν ε, τις ε, εταιρείε, άλλε όχι. Η Γερμανία και η Ιταλία, για να δώσω ένα παράδειγμα, και αυτό δημιουργεί στρέβλωση στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να διορθωθεί. Ο μόνο τρόπο να διορθωθεί είναι με τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για αυτέ τι αποζημιώσει. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πολύ, Γέρση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπινκόφσκα. Ε, Καταρχά, θα ήθελα να σα πω ότι ελπίζω και σε δύο εβδομάδε από τώρα να είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούμε. Διότι μόνο όλοι μαζί και 28 μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Κίνα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε όπως καταστρέφονται ολόκληρες κοινότητες όταν ε, καταστρέφονται οι βιομηχανίες που τις στηρίζουν η αλυσίδα διανομής έχει υποφέρει και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Τώρα, σε σχέση με την Κίνα, βλέπουμε ότι έχουν τελείως διαφορετικά πρότυπα. Ε, εκεί κυριαρχεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ε, αλλά δεν είναι μόνο οι τομείς που αναφέρεται. Και η κεραμοποιία και η αλλουργία υποφέρει εξαιτία των αθέμητων πρακτικών της Κίνας. Αυτό έχει κοστίσει εκα, ε, χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Καθήκον μας λοιπόν είναι να προστατεύσουμε αυτές τις θέσει απασχόλησης και τις κοινότητές μας. Τώρα, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, Φαίνεται πως χρειάζεται δράση γι' αυτό και χρειάζεται δράση η οποία θα ωφελήσει τους φτωχότερους. Είναι σκανδαλώδες το ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Χρειάζεται ανακαίνιση κατοικιών ε, στις οποίες ε, κατοικούν σε απόλυτα άσχημες συνθήκες άνθρωποι και αυτό είναι απίστευτο και απαράδεκτο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, χρειάζεται μια κοινή βιομηχανική πολιτική. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο αρμοδιότητα δύο επιτροπών, της δικής μας και της επιτροπή Πολιτισμού ε, και δεν πρέπει μόνο να μείνουμε στα λόγια, πρέπει να γίνουν πράξεις, πρέπει να προστατεύσουμε την ε, αλυσίδα εφοδιασμού και διανομή για να προστατεύσουμε του πολίτε μα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Η Κίνα δεν είναι οικονομία της αγοράς. Μόλις το είπατε ή το επαναλάβατε. Ωστόσο, μας ε, λέτε ότι είναι δύσκολη η συζήτηση ε, στις η Ιουλίου στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Αλλά εκπλήσωμε εκπλήσωμε. γιατί είναι πολύ καθυστερημένη, έρχεται πολύ καθυστερημένα αυτή η συζήτηση. 23 Ιουλίου έχουν ήδη ξεκινήσει ε, οι διακοπές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένως δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε παρά πριν το Σεπτέμβρη. Μήπω είναι παγίδα αυτή η ημερομηνία, παγίδα που κάποιοι συνάδελφοί σας ε, θέλουν να βάλουν μια τρικλοποδιά α πούμε στους βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι μόνο σε εμά. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη ομόφωνα ε, το ε, ε, ε, Συνδικάτο ενδυστριών που εκπροσωπεί πολλούς εργαζόμενους από πολλούς βιομηχανικούς κλάδους εκφράστηκε επ αυτού του θέματος καλώντας το, την Κομισιόν να μην δώσει αυτό το καθεστώς στην Κίνα. όσον αφορά τώρα το ETS και μια και το μιλάμε, εγώ σαν παλαιός εργάτης χαλιβουργίας σας λέω ότι είναι καλό πράγμα αυτό το σύστημα ε, ανταλλαγής εκπομπών ε, και για, τους, ε, για το κλίμα και για τον πλανήτη αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα είναι καλό και θα έχει αποτέλεσμα εάν ισχύσει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο και θα πρέπει όλοι και οι επίτροποι να καταλάβουν πραγματικά ότι η Ευρώπη δεν είναι μοναχή της στη μέση του κόσμου. Νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε ε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε, να πολεμήσουμε αυτήν την τιμή του χάλιβα ε, που προέρχεται από την ε, Κίνα. 37 εκατομμύρια τόνοι ε, έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν ε, κοστίσει 10 ευρώ το ε, διοξίδιο του άνθρακα τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε, να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία χωρίς επιπλέον κόστος. Βλέπουμε ότι οι επίτροποι σιωπούν ε, και αύριο θα πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτή την κατάσταση, αυτή την ένοχη σιωπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιος ζητά το λόγο. Όχι. Επομένως, ε, κυρία Επίτροπε, παρακαλώ να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ανά ομάδες. Και εάν δεν σας απαντήσω τώρα θα σας απαντήσω γραπτά. Όσον αφορά αυτό το 20% ε, ή μάλλον το ε, ποσοστό της βιομηχανίας ε, στην οικονομία μας. Ναι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να επιτύχουμε αυτό το 20% αλλά νομίζω ότι η κυρία Γρυπηδίδη απάντησε στην ε, ε, ερώτηση εν μέρη τουλάχιστον η βιομηχανία ε, ή πρέπει να πούμε ότι επηρεάζεται ή εξαρτάται από άλλα στοιχεία όπως είναι οι υπηρεσίες, όπως είναι η γραφειοκρατία κτλ. Επομένως υπάρχουν για τα θέματα της βιομηχανίας, της καθαρής βιομηχανίας κλπ. και άλλα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν. Μακροπρόθεσμα επενδύουμε ή ε, αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά πιστεύω ότι στην βιομηχανική μας στρατηγική μπορείτε να βρείτε την πλήρη απάντηση την στρατηγική ε, που θα δημοσιοποιήσουμε τον επόμενο χρόνο, γιατί εκεί ακριβώς ε, θα αναφέρεται η διασύνδεση των υπηρεσιών. Ε, ε, γιατί ας πούμε έχουμε περιπτώσεις όπου, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου 70% ε, του τζίρου φορά τις υπηρεσίες. Του χρόνου λοιπόν η σαφής απάντηση όταν θα δημοσιοποιηθεί η στρατηγική. Αλλά να υπενθυμίσω ότι δεν μιλάμε μονάχα για την βιομηχανία, την παραγωγή, δηλαδή αυτή καθεαυτή παραγωγή του προϊόντος. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Ενέργεια. Πολλές ερωτήσεις για την ενέργεια. Πρέπει να πω ότι ούτε εγώ ούτε ε, η Επιτροπή θα δεχτούμε αύξηση τιμών. Δεύτερον, αυτός είναι και ο στόχος, ο κύριος στόχος ε, της ε, αγοράς ενέργειας και της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Εμείς δεν θέλουμε την ενέργεια η οποία θα αντιμάχεται την βιομηχανική ανάπτυξη γιατί αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε, αλλά ούτε είναι δυνατόν να αντέξουμε τη ζωή σε μια κοινωνία η οποία δεν σέβεται τους ε, ε, στόχους ε, για το κλίμα. Είναι υψηλή οι στόχοι και οι υψηλές αποφάσεις αυτές που λαμβάνονται στο Συμβούλιο και που μετά περνούν από την Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το θέμα αυτό βρίσκεται στους συνομοθέτες. Εμείς οπωσδήποτε θα συμβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο, άλλωστε το έχουμε ξανακάνει. Στις προηγούμενες προτάσεις της Κομισιόν, τις προτάσεις δηλαδή που στέλνουμε και στο ε, Συμβούλιο υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές. Ε, ξέρω ότι οι αποφάσεις που πήραμε και οι προτάσεις που κάνουμε δεν αρκούν στην βιομηχανία κυρίως για τις πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και γι' αυτό ακριβώς προτιθέμεθα να επανασχεδιάσουμε και να τροποποιήσουμε το σύστημα ETS. Σας το είπα ξανά ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη βιομηχανία αλλά ούτε μπορεί ε, να εγκαταλείψει και τις ε, φιλοδοξίες που έχουμε σε άλλους τομείς όπως είναι ας πούμε το κλίμα γιατί αλλάζει ο κόσμος, άλλωστε και εγώ έχω αλλάξει ε, λίγο, έχω μετακινηθεί όσον αφορά τις θέσεις μου. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να διανύσουμε αυτήν την περίοδο που θα κρατήσει αρκετά χρόνια χρόνια έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα πράγματα πάνε καλά. Βεβαίω θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την ε, ε, ενεργειακή ε, ασφάλεια. Όλα αυτά τα στοιχεία θα περιληφθούν στις απαντήσεις μας και στις συζητήσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Ε, ελεύθερες ποσοστώσεις ε, ETS δωρεάν ε, λοιπόν δικαιώματα αυτό βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου έτσι ώστε να δοθούν ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια της αγοράς. θα είναι πολύ δύσκολο μια τέτοια ιδέα να περάσει από το Συμβούλιο. Κίνα και χάλιβας. Ή μάλλον όχι να πω κάτι άλλο, αναφερθήκατε σε άλλους τομείς ε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ε, το ανταγωνισμό. Ναι, βεβαίως ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας έτσι ώστε να προστατέψουμε τους ε, παραγωγούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός άμυνας και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε και πιο ενεργητικά εργαλεία προστασίας του εμπορίου. Ξέρω ότι δεν έχουν γίνει αρκετά μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά έχει υπάρξει και μια εμπλοκή στο Συμβούλιο. Μιλούσα προημερών με την Ολλανδική Προεδρία ε, γιατί υπάρχουν θέματα που ε, ούτε συνεργαζόμενοι μαζί τους μπορούμε να τα προωθήσουμε γιατί πολλά κράτη-μέλη αντιστέκονται ακόμα και ε, κράτη-μέλη τα οποία φαίνονται ιδιαιτέρως να υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Ε, και η Κομισιόν και το, Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ε, προσπαθεί να προωθήσει τα πράγματα, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλά ε, κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δεν ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο σκέψης μας. Εμείς προσπαθήσαμε να ε, στους τελευταίους έξι μήνες να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ε, και έχουμε δουλέψει πολύ και με τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα εμπορίου, αλλά δεν προχωράνε τα πράγματα όπως θέλαμε. Τώρα Κίνα και ε, το καθεστώς της δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις σχετικά με το κατά πόσον η Κίνα θα θεωρηθεί κράτος οικονομίας αγοράς. Ε, η προσωπική μου άποψη ε, είναι ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και οπωσδήποτε θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια ε, πιο εξεζητημένη ας πούμε λύση. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί γιατί σύντομα θα υποβληθούν προτάσεις από την Κομισιόν. Είναι γνωστές ε, οι απόψεις μου για το θέμα. Ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμό ε, τους επόμενους, τις επόμενες εβδομάδες και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει αυτός ο συμβιβασμός. Όσον αφορά το EFSI και το πρόγραμμα COSPA. Ήδη, ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα του Ταμείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιομηχανικά ε, προγράμματα και το έχω ε, πει και το έχω τονίσει επανειλημμένα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο υποδομές βιομηχανικές αλλά ε, και συγκεκριμένα προγράμματα. Τα κράτη υποβάλλουν προτάσεις, όχι πάρα πολλές, αλλά πάντως υποβάλλονται και κάποιες βιομηχανικές προτάσεις. Ε, άλλωστε, στο Ταμείο υπάρχει και αυτό το στοιχείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, επομένως ανοίγει μια τεράστια ευκαιρία για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μέχρι τώρα οι συμβάσεις ε, που έχουν υπογραφεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, δεν είναι πάρα πολλές, ε, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία. Στα θέματα των υποδομών τα πράγματα προχωράνε πιο γρήγορα. Όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, Δεν είμαι πλήρως ικανοποιημένη από τον τρόπο λειτουργία του κόσμου, το οποίο είναι πολύ καλό εργαλείο με 2,8 δις είναι ένα ένα καλό εργαλείο χρηματοδότησης, ε, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι του χρόνου. Ε, δεν μπορώ να πω ότι με προβληματίζει ο τρόπος, με τον, ο, η ροή του χρήματος, αλλά τα κύρια κριτήρια ε, και οι αποδέκτες των πόρων ίσως είναι στοιχεία πιο προβληματικά ε, ίσως ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, σημασία και στο ψηφιακό κομμάτι της αγοράς. Θα το δούμε. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους και την βιομηχανία σχετική με τους σιδηροδρόμους, αυτά που είπε ο κ. Βέρνερ είναι πολύ σημαντικά. κυρία Βέρνερ. Αυτές ε, οι εταιρικέ σχέσεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι κάτι θετικό και πιστεύουμε ότι είναι τμήμα της απάντησης. Ε, του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό όντως μπορεί να ε, υπάρξει καινοτομία ε, και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να είμαστε απολύτως ε, ανοιχτοί. Άλλωστε η Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια κατά αυτή την έννοια τοποθετήθηκε. Πιστεύουμε ότι και η πρωτοβουλία υπέρ του σιδηροδρόμου μπορεί να αποτελέσει, να δώσει μια σημαντική όθηση. Τι άλλο όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα. Η πρόταση βασίζεται ούτως ή άλλως στις βέλτιστες ε, πρακτικές των κρατών μελών. Τώρα η συζήτηση βρίσκεται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, στην, ε, στο τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 9ης Ιουνίου συζητήθηκε το θέμα αυτό. Βλέπουμε τις εθνικές νομοθεσίες, αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν είναι αρκετές. Εμείς προσπαθήσαμε όλα τα σημαντικά στοιχεία να τα βάλουμε σε μία δέσμη. Ξέρω ότι οι κυνηγοί έχουν διαφορετική άποψη ε, και κάποιες άλλες ομάδες, αλλά πραγματικά σας, ε, ε, σας ζητώ, σας κάνω έκκληση, απευθύνω έκκληση, έτσι ώστε να προωθήσετε αυτή τη δέσμη. Α, και κάτι άλλο. Benchmark για το ε, ETS. Κύριε Νίκα, όπως είπα και προηγουμένως, ε, ενεργούμε και δραστηριοποιούμεθα και εγώ ιδιαίτερος ε, για το ETS και για μία ακόμα φορά πρέπει να πω κάτι που είπα επανειλημμένα είναι εύκολο να επιτεθεί κανείς στην Κομισιόν για τις προτάσεις που κάνει. Αλλά οι πρώτες προτάσεις και οι πρώτες γενικές κατευθύνσεις λαμβάνονται σε υψηλό επίπεδο στο Συμβούλιο. Ακούω παράπονα από τους ε, Υπουργούς Βιομηχανίας ε, ή τους Υπουργούς Οικονομικών για το ETS. Αλλά έχουμε στοιχεία όπως είναι ας πούμε οι συμφωνίες για το κλίμα όπως το Παρίσι ε, και αυτές λαμβάνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Η Κομισιόν στην ουσία εκτελεί τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι άδικο να επιτίθεται κανείς ε, στην Κομισιόν έστω και εάν ε, εγώ πάντα βρίσκομαι στο πλευρό της βιομηχανίας, αλλά πρέπει να πω και να ξαναπώ ότι αλλάζει ο κόσμος και σε 20-30 χρόνια η βιομηχανία μας θα είναι εντελώς διαφορετική. Με ρωτήσατε και για τον άνθρακα. Πιστεύω ότι μαζί με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουλέψουμε, να βρούμε στρατηγικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να δώσουμε διαφορετική μορφή στην βιομηχανία μας τα επόμενα χρόνια. Έχουμε τώρα και το θέμα της ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας και ο καθένας προσπαθεί από την δικιά του ε, πλευρά για μένα. Η βιομηχανία είναι η κύρια προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις και τα σχόλιά μας. Και Ελπίζω να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την επόμενη συνάντησή μας για το φθινόπωρο, διότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το 2017, όποτε και θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την ανταλλαγή απόψεων. Καλή συνέχεια κυρία Πίτροπε. Έχετε πολλά να κάνετε, πολλές δραστηριότητες για το 2016. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Και ε, να μας ξανάρθετε τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Um. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες μου και κύριοι, επόμενο θέμα στην ημέρα διάταξη. Πάρα πολύ σημαντικό. Προτεραιότητες της ΣΥΤΡΕ στον προπολογισμό του 2017. Πριν από λίγο ανέφερα ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε από τώρα για το 2017 το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου εν γέννη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 και στο διαρθρωμένο μας διάλογο με τους επιτρόπους. Πλην όμως, τώρα έχουμε τον προπολογισμό για το 2017 που θα είναι επίσης πολύ σημαντικός και έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιάννη Γκάια για αυτό το θέμα. Που είναι συγητής της Επιτροπής Προπολογισμών. For είναι συγητής του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. Dear colleagues, if I Uh, uh, Έλεγα λοιπόν ότι είναι εδώ ο κύριος Γκάιε. Θέλει το λόγο η κυρία Τόγια προηγουμένως. Ορίστε. Μία γενική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να διακόψω τη σειρά των εργασιών. Δεν είναι εδώ ο Σνάρφρου Γκάγερ. Όταν θα τελειώσει το σημείο αυτό, μετά τα λέω εγώ. Α, νάτος, εδώ είναι. Όταν τελειώσει, όταν τελειώσει θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα. Αλλά φίλε και Ένα λεπτό λοιπόν, Σαν Γκάγερ, να πω κάτι στον Πρόεδρο. Μερικές φορές ε, ε, πολύ συχνά μάλιστα δεν ε, απαντώνται οι ερωτήσεις. Ίσως ε, είτε εγώ δεν έκανα καλά την ερώτηση είτε δεν κατάλαβε η Επίτροπος γιατί δεν μου απήντησε. Κάποια στιγμή ή τα μέλη της Κομισιόν, οι Επίτροποι, οι εμπειρογνώμονες όταν έρχονται εδώ θα πρέπει να απαντάνε ναι, στις ερωτήσεις μας ή εάν δεν κατάλαβαν την ερώτηση, ας πούμε η κυρία Επίτροπος δεν κατάλαβε Βέλγιο. Θα έπρεπε να μου είχε πει η κυρία Τόγια, δεν κατάλαβα την ερώτησή σα, να μου την ξανακάνετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ε, γιατί τι να σα πω, ούτε σε εσά απήντησε, ούτε σε μένα. Η Επίτροπο απήντησε εκεί που ήθελε, όπω ήθελε. Ε, δηλαδή, πραγματικά αυτή η υπεκφυγή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Εδώ που τα λέμε δεν θυμάμαι όλες τις ερωτήσεις που έγιναν, γι' αυτό μου είναι δύσκολο να τοποθετηθώ για το αν απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις ή όχι. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι ολοφάνερο ότι στις επόμενες συναντήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά ε, την τελευταία τοποθέτηση της ε, κυρίας Επιτρόπους θα σας ρωτήσω αν θέλετε να επαναλάβετε κάποια ερώτηση γιατί δεν απαντήθηκε και μετά θα είναι σαφές για μένα τι έχει γίνει και τι όχι. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι σαφές. Καμιά φορά ε, ζητάτε το λόγο, λέτε κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, σας δίνω το λόγο μετά. Μετά την τοποθέτηση του Επιτρόπου. Αυτή τη φορά δεν ζήτησε κανείς το λόγο μετά τα τελευταία σχόλια της Επιτρόπου. Γι' αυτό λοιπόν δεν αντέδρασα. Στο μέλλον θα σας ρωτάω. Τα λέω, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχουν ε, αναπάντητες ερωτήσεις, όχι νέες ερωτήσεις, αναπάντητες. Γιατί αν κάνουμε και άλλες ερωτήσεις θα τελειώσουμε ούτε σε δύο ώρες. Θα ρωτώ λοιπόν και από εδώ και στο εξής έτσι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια, πολύ καλή πρόταση κάνετε. Θα την ακολουθήσουμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχετε το θάρρος να το ρωτήσετε ίδια. Μάλιστα. Όχι, ε, απλώς έχω καλή αγωγή. Budget. Καλώς. Είμαστε όμως στο προπολογισμό τώρα στο σημείο 16. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε για την εντολή ε, της Ήτρε και είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. να ξέρουμε ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα, να έχουμε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Και ξέρουμε, ε, αν ξέρουμε ποια είναι τα θέματα που μας ε, ενδιαφέρουν, χρειαζόμαστε και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου θα καταθέσει το σχέδιο προϋπολογισμού ένα μήνα αργότερα από την αρχικά αναμενόμενη ημερομηνία. Η δική μας νέα προθεσμία για τις τροπολογίες, για τις γραμμές του προπολογισμού, θα είναι η 5η Ιουλίου πλέον, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αναβάλαμε και εμείς και τη συζήτηση και την ε, προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Η δε ψηφοφορία πάντα στην Ήτρε θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξή, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητώ συγγνώμη που θα το πω, όλες οι τροπολογίες πρέπει να είναι στα αγγλικά. Λυπάμαι. Δεν θα πρέπει να λυπάμαι. Εν πάση περιπτώσει θα είναι κάπως δύσκολο φαντάζομαι για εσάς να τις συντάξετε στα αγγλικά. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή από όλε τι γλώσσες στα αγγλικά. Γιατί για αυτό το λόγο χρειάζονται τρεις εβδομάδες μέσα σε λίγες μέρες δεν προλαβαίνουμε. Ανάμεσα στην κατάθεση της προθεσμίας, μάλλον στη λήξη προθεσμίας για την κατάθεση των τροπολογιών και την ψηφοφορία δεν μεσολαβεί αρκετό διάστημα και γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε τις τροπολογίες σας στα αγγλικά, στις 12 το μεσημέρι, μέχρι, λοιπόν, εκείνη την ώρα της 5ης Ιουλίου. Χρόνο πολύ δεν έχουμε. Στις 13 Ιουλίου είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα τα πει σίγουρα και ο συγγητής μας. Γενικές συστάσεις, η γνωμοδότησή μας θα συμπεριληφθεί σε αυτές τις συστάσεις του εισηγητού και της Επιτροπής Προπολογισμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν και οι δικές μας προτεραιότητες στο φάκελο αυτό. Γιατί να θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον ε, εισηγητή μας να τα συμπεριλάβει στις δικές του συστάσεις. Ε, γιατί την πρώτη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου. Το λόγο ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Πολύ ωραία συνοψίσατε την κατάσταση και με μεγάλη ακρίβεια. Κανονικά τώρα θα έπρεπε εδώ και τρεις εβδομάδες να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 και με την αντιπαράθεση αυτή με την εξέταση του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε κατά τέσσερις εβδομάδες την επίσημη κατάθεση με επίσημη δικαιολογία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπεσε έξω στο κόστος της προσφυγικής πολιτικής, δεν έχει ακόμα τελειώσει τους υπολογισμούς και στις 25 Ιουνίου θα τα έχει κάνει όλα αυτά. Καμία σχέση με τον προϋπολογισμό. Καμία σχέση και εντελώς τυχαία είναι μετά το βρετανικό δημοψήφισμα όλο αυτό. Όλα αυτά είναι εικασίες και είναι τρομερά άδικο αυτό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά εμπαρόδο το λέω. Εντελώ κατά τύχη το έχουν βάλει μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έχει γίνει στο μεταξύ. Από τα τέλη Απριλίου και την απόφαση της Ολομέλειας υπάρχει σαφή θέση για τις δικές μας προσδοκίες. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, λεγόμενες guidelines ήδη οι λιμένες αποφάσεις για τους μεγάλους προσανατολισμούς και ελπίζω να έχουμε μεγάλη ε, υποστήριξη, γιατί πέρασε και με μεγάλη πλειοψηφία. Και ελπίζω να μας διέπουν αυτές οι αρχές ε, μέχρι ε, να αποφασιστεί ο προπολογισμό που ελπίζω να μην αργήσει πάρα πολύ φέτο. Θέλω να θυμίσω το εξή. Πώ έχει η κατάσταση. Ο προπολογισμό του 2016, ο τρέχον τώρα, για το παρόν οικονομικό έτος, έχει τεράστιες προκλήσεις. Αρκεί να σας αναφέρω τις μεγάλες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται με την προσφυγική κρίση και πιέζουν τις κατηγορίες 4 που είναι η εξωτερική πολιτική καταπολέμηση των αιτίων της προσφυγιάς και κατηγορία 3 που μεταξύ άλλων εσωτερική πολιτική που έχει να κάνει με την υποδοχή στα κράτη-μέλη για να ε, βοηθήσουμε λίγο τα κράτη-μέλη και να ελαφρυνθεί ο προπολογισμό του τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί πλήρως, δεν υπάρχει ε, κανένα περιθώριο ανάμεσα στο ανώτατο όριο που ορίζει το πλαίσιο των, ε, δημοσιονομικών προοπτικών και τον προπολογισμό του 2016. Οι κρίσει αυτές δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται όλες. Μακάρι να μπορούσα να είμαι πιο αισιόδοξο ε, για το μέλλον από ό,τι είμαι. Δυστυχώ δεν βλέπουμε καμία ένδειξη ότι οι αιτίες ε, της προσφυγικής κρίσης ε, θα εκλείψουν ή ότι θα καταφέρει η πολιτική να εξαλείψει αυτές τις αιτίε, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των προκλήσεων που είχαμε φέτος θα συνεχιστούν και το 2017 και θα μας συνοδεύουν και το 2017 με ε, την αντίστοιχη επιβάρυνση του προπολογισμού. Έχουμε και την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, δεν έχει ξεπεραστεί απολύτως και πλήρωσε όλα τα κράτη-μέλη. Και σε σχέση με αυτό θέλω να πω και πώς έχει το πολιτικό κλίμα και το περιβάλλον στην ε, θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει, επέβαλε έκτακτα οικονομικά εργαλεία και μέσα. Διαφωνούμε με το Συμβούλιο και δεν τα έχουμε βρει ακόμα εάν και κατά πόσο αυτά τα έκτακτα μέσα θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προπολογισμού. Αυτό λέει η Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου. Η περίφημη διατύπωση που είχαμε σε αυτό το ψήφισμα την πάγια ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να κινούνται πάνω και πέρα από το ανώτατο όριο, above and beyond. Ενώ το ε, Συμβούλιο το βλέπει ακριβώς αντίθετο, εντός των ορίων. Ναι, αλλά ο προπολογισμό ε, ήδη θα είχε εκραγεί αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε επιβάλει αυτά τα έκτακτα οικονομικά μέσα θα μας είχε ξεφύγει τελείως. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο που πρέπει να δούμε σε σχέση με τον προπολογισμό και το δεύτερο είναι κάτι που έχει να κάνει περισσότερο με την καθημερινή δουλειά της Επιτροπής εδώ, ΙΤΡΕ. Θα πρέπει να βρούμε χρήματα για να ε, καλύψουμε τις εγγυήσεις του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. 3,38 ε, δις έχουμε κινητοποιήσει. Υπάρχει κάποιο περιθώριο μέχρι τα 8 δις που πρέπει να κινητοποιηθούν. Και αυτά θα πρέπει να βρεθούν από τον επόμενο προπολογισμό. Και ακόμα δεν έχω πει τίποτα για επιπλέον οικονομικές ε, ανάγκες από τη διευκόλυνση για την Τουρκία και κάτι άλλα ψηλά που μπορεί να μας προκύψουν. Άρα, κατά την άποψή μου, είναι όλο και προφανέστερο ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει αυτό το καιρό ε, είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να πάει καλά αν δεν έχουμε κανένα ε, απρόπτο. Το 2013 όλα αυτά φαινόντουσαν πάρα πολύ ωραία γιατί δεν ξέραμε τι θα μας προκύψει. Έκτοτε έχουμε συνεχιζόμενες διαρκείς κρίσεις και τεράστιες απαιτήσει ε, που ε, πραγματικά το πλαίσιο αυτό έχει τόσο πολύ ξεχυλωθεί που κινδυνεύει να σπάσει. Επιπλέον, έχουμε και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κάθε φορά που θέλουμε να τονίζουμε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και θα πρέπει να συνδέονται τα κονδύλια με τις οικονομικές εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις που γίνονται. Δηλαδή, έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομική προοπτική. Τελευταία ήταν το φθινόπωρο του 2015. Έχουμε αιτήσει έκθεση ανάπτυξης. Έχουμε ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και νομίζω καλά θα κάναμε να αναπτύξουμε περισσότερες συνέργειες μεταξύ του προπολογισμού και όλων αυτών των οικονομικών εργαλείων, εργαλείων οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να αποκτήσουμε περισσότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν μιλάω για τις συστάσεις αναχώρα τώρα, ε, από το οικονομικό ευρωπαϊκό εξάμεινο, ότι θα έπρεπε ένα προς ένα να υιοθετηθούν, γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο το κοινοβούλιο το ίδιο θα καταδίκαζε το εαυτό του σε αιώνια σιωπή. Αλλά κάπως να τα λαμβάνουμε υπόψη και έχουν αποφασιστεί και από τις κατευθυντήριες γραμμές του Επιπλέον, τα προβλήματα αυτά που αναλαμβάνω δεν έχουν εξαφανιστεί, ούτε πρόκειται. Υπάρχει στρατηγική ορίζον 2020. Μάλλον όχι, διορθώνει ο μιλητής. Ευρώπη 2020. Παράδειγμα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, η οποία θα πρέπει να μεταξελιχθεί, η καταπολέμηση της φτώχειας, που είναι στόχος δηλωμένος στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, ιδιαίτερα για την παιδική φτώχεια. Θα πρέπει να πιάσει τόπο. Κάτι το οποίο χαλάρωσε κάπως είναι η κατάσταση της πληρωμές, γιατί υπήρξαν ε, μετρητά. Στο τελευταίο πλαίσιο είχαμε ένα τσουνάμι ε, ε υπερημερών πληρωμών, ανεξόφλητων ε, λογαριασμών που κάπως έχουν καλυφθεί γιατί έχουμε νέο χρήμα φρέσκο τώρα με τις νέες προοπτικές αλλά το χάσμα από τις την ανάληψη υποχρεώσεων ε, είναι 907 ε, δις και 50 δις υποχρεώσεις πληρωμών. Υπάρχουν κάποια πολιτικά σχέδια που έχουν προγραμματιστεί και έργα που είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ε, αν δούμε τι κάνει το Συμβούλιο, είναι πραγματικά ε, επιπόλαιο. Μπορεί το 2016-2017 αυτά τα ράλ τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, το rest αλικείται ε, όπως ε, λέγεται αυτό στη γλώσσα των ειδικών, θα έχουμε πρόβλημα. Ο πρόεδρος Ζακόπτη, θα πρέπει να έχουμε ένα προπολογισμό λοιπόν αντίστοιχο και περιμένω με χαρά τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αρχίσουμε με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, η οποία, όπως είπα, ψηφίστηκε σήμερα το πρωί. Οπότε θα ήθελα να αναφέρω τα πιο σημαντικά σημεία της γνωμοδότησης αυτής. Ε, καταρχάς, θα θέλαμε ο προπολογισμό του 2017 να διευκολύνει την ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη, έξυπνη και βασισμένη στη γνώση. Αυτό συνεπάγεται και ουσιαστική χρηματοδότηση. Και ίσως η καλύτερη πρόταση είναι τα πολιετή προγράμματα, όπως το κόσμο ορίζοντας 2020 κτλ. Αυτά είναι απολύτως αναγκαία και όντως έχουν εντοπιστεί προβλήματα από καιρό σε καιρό στη χρηματοδότησή τους. Επίσης, ζητάμε διόρθωση των γραμμών προπολογισμού για τον ορίζοντα 2020 και το συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να επιμείνουμε πάνω του. Ε, ενίσα, Ενίσα, S ε, για security, ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ε, η ψηφιακή ενιαία αγορά και η ψηφιακή ένωση είναι κάτι που παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά και θεωρούμε πολύ σημαντικό. Όλο ένα και σημαντικότερο. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στον χώρο της ενέργειας. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να ε, επιτευχθούν οι στόχοι της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Πολύ σημαντικό. Διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών, παρόχων, συνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα και για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό. Επίσης, άσερ, η ε, υπηρεσία ρυθμιστικών αρχών ενέργειας θεωρούμε επίσης πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Επαρκής πόρη είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της ΆΣΕΡ. Και έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στα προγράμματα ITER. Θα χρειαστεί να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις στο προσεχές μέλλον. Γι' αυτό και θα χρειαστεί μια διαβούλευση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Αυτό θα γίνει σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Δεν πρέπει όμως ε, σε καμία περίπτωση να το παραμελήσουμε. Τώρα, η κυρία Επίτροπος Γεωργίευα, αντιπρόεδρος Επιτροπής, είπε ότι υπάρχει προϋπολογισμός ε, για ε, το θεματολόγιο αποτελεσμάτων. Τι σημαίνει αυτό για την πολιτική της Επιτροπής μας. Πολλά. Χρειάζεται όμως να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό. Και οι συνέργειες είναι πολύ σημαντικές. Συνέργειες ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και όλους ε, τους ε, άλλους ε, διαθέσιμους πόρους του προπολογισμού για την καινοτομία, για την ανάπτυξη. Συνέργειες που θα συνδέονται με τις πρωτοβουλίες για ε, έξυπνη εξειδίκευση. Και αυτό θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, βασικό στοιχείο του προπολογισμού μας. Αυτά λοιπόν ε, ε, ως προτεραιότητες που ψηφίστηκαν σήμερα από την Επιτροπή μας. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στα σχόλια των μελών της Επιτροπής. Ποιος θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο και θεωρεί πως θα είναι σημαντικό σχόλιο για τον εισηγητή. Κυρία Κάπελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Γκάιερ για αυτά τα λόγια του, για αυτές τις ρεαλιστικές προβλέψεις για το 2016 και τώρα για τον προπολογισμό του 2017 και για το τι αναμένουμε. Πιστεύω πως είναι πολύ καλό να είμαστε πραγματιστές, να είμαστε ρεαλιστές για να δούμε πώς θα διηγηθούμε στον στόχο. Ε, και όπως είπατε και εσείς δεν πρέπει να βάζουμε στόχους που θα επιτευχθούν μόνο όταν όλα θα πάνε καλά, πρέπει να προβλέπουμε τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν ε, κύριε Πρόεδρε, το είπατε και εσείς, το είπε και ο κύριος Γκάιερ, ότι οι ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχουν ε, μειωθεί. Έχουν μειωθεί και αν δει κανεί όλα τα έργα τα οποία ε, πρέπει να γίνουν και συμπεριλαμβάνονται στον προπολογισμό της ενέργειας, ψηφιοποίηση, ενεργειακά θέματα, το ΙΤΕΡ. Τότε, αν δει κανεί όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι ε, αναλήψεις υποχρεώσεων ε, δεν μπορούν να μειωθούν αν θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αναπτύξουμε υποδομές για την Ενεργειακή Ένωση, για να κάνουμε όλα αυτά που είναι αναγκαία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πράγματι οι προκλήσεις όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό είναι τεράστιες και η Επιτροπή μας έδειξε μεγάλο ε, θάρρος σήμερα ψηφίζοντας την διαπραγματευτική εντολή για τον τριμερή διάλογο. Έδειξε προς τα που θέλει να πάει, έδειξε πως γνωρίζει ποιο είναι το κόστος της αποτυχίας, έδειξε πως είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και πως ε, χρειάζεται εσεί στην Επιτροπή του Προπολογισμού να καταπιαστείτε με αυτό το δύσκολο θέμα, με τη δύσκολη πρόσκληση και να δώσετε απαντήσει. Πρέπει να τις βρείτε αυτές τις απαντήσεις και σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαραγκάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Ο κύριος Γκαγιέρε ε, αναφέρθηκε προηγουμένως στις ε, καθυστερήσεις ε, όσον αφορά τα έγγραφα της, τα πρώτα της Κομισιόν και την σχέση αυτής της καθυστέρησης με το δημοψήφισμα στην Βρετανία ε, ε, έστω και αν ε, κάποιος θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσει κάπως την εικόνα. Αυτό βεβαίως είναι το άκρονάο των, της θεσμικής χρήσης κάποιων στοιχείων. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στο Κοινοβούλιο, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια δεν νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ θετικά όσον αφορά και το δημοψήφισμα. Θα δούμε θα δούμε εάν ε, ε, η σιωπή μας ήταν υπερβολική και αν ε, ενδεχομένως η υπερβολική προσοχή μας έδωσε τα αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τον Brexit. Κύριε Γκάγερ, άκουσα αυτά που είπατε και πραγματικά σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε στην Επιτροπή των Οικονομικών. Μονάχα να πω δύο λόγια ε, την επόμενη χρονιά θα είναι η πρώτη χρονιά μετά την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ε, ίσως και ενδεχομένως μόνο και για αυτό τον επίσημο ε, λόγο, ε, θα πρέπει κάποια πράγματα να φανούν σαφέστερα στον επόμενο προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Δεν είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ έντονες τον, τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Τώρα είναι ε, ίσως ε, ε, πιθανό ή εύκολο να υποπέσουμε στον κίνδυνο να έχουμε υπερβολικά αιτήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι ορισμένα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρώτον, energy transition. Αυτή η ιδέα πρέπει να είναι σαφής και να προχωρήσει. Δεύτερον, ε, στόχοι 2020 πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην καινοτομία ε, ή εν πάση περιπτώσει πολιτική, ε, βιομηχανική πολιτική σε σχέση με την καινοτομία έτσι ώστε να έχουμε έρευνα και, και καινοτομία σωστά. Επίσης ένα ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό ή που θα ανοίξει με αυτήν την συζήτηση, δηλαδή ε, η αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού ε, ε, πλαισίου και το θέμα των runs to loans. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει καθαρά. Άλλο είναι το grants, άλλο είναι τα loans θα πρέπει να βρεθούν συνέργειες, σημαντική λέξη η οποία μπορεί να είναι της μόδας αλλά είναι πολύ σημαντική και βεβαίως αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην συζήτηση που τώρα θα ανοίξει ε, πραγματικά την σχέση ανάμεσα σε ανταγωνιστικότητα και ε, συνέχεια. Θα πρέπει να είμαστε ε, φιλόδοξοι, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια νέα ισορροπία, αλλά όχι χαλώντας τον προϋπολογισμό και προσπαθώντας να βρούμε ένα νέο νέο υπόδειγμα το οποίο δήθεν θα μας βγάλει από όλα τα προβλήματα. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι καλό. Και κάτι τελευταίο, ή μάλλον πρώτο τελευταίο, ε, το COP21 Πρέπει να πω ότι η ομάδα καταψήφισε ε, την γνωμοδότηση, έστω και αν ε, οι συμβιβασμοί έγιναν δεκτοί. Καταψηφίσαμε γιατί στην περίπτωση του ΙΤΕΡ δεν ε, ταυτίζεται με την αρχή της προσοχής που είχε υπογραμμιστεί και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιλ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω κύριο Γκάιερ. Είναι το καλύτερο να είμαστε ανοιχτοί όταν συζητάμε για οικονομικά θέματα και όταν λέμε ότι έχουμε δαπανίσει 50 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσο έπρεπε, τότε ε, είναι καλό να το ακούμε και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ε, διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά η απάντηση σε αυτό δεν είναι ε, ναι, η Επιτροπή Προϋπολογισμού πρέπει να σκεφτεί για το πώς θα εξοικονομήσει πόρους ή πώς θα κάνει περικοπές. Όχι, χρειάζεται να σκεφτούμε σε ε, μεγαλύτερη κλίμακα, να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα έτσι ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Διαφορετικά θα πέφτουμε όλο ένα και πιο μέσα στη μαύρη τρύπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλοάγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φτάσαμε ε, να συζητούμε τον προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο και από την άποψή μας αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Μπορούμε να έχουμε και να προτείνουμε πολλούς στόχους για τον επόμενο ε, χρόνο, αλλά αν η χρηματοδότηση δεν ακολουθήσει τότε θα είναι καινό γράμμα. Ε, η συζήτηση για τον προπολογισμό πάντω είναι σημαντικό, όχι μόνο όσον αφορά τι δαπάνε, αλλά και όσον αφορά τα έσοδα. Κατά αυτή την έννοια εμείς λέμε ε, ότι θα πρέπει να ε, αυξηθεί ο προϋπολογισμός ε, αλλά να είναι πιο ευέλικτος έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις κρίσεων όπως ας πούμε αυτή των προσφύγων. Και όσον αφορά τα έσοδα πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο δίκαιο και πιο προοδευτικό σύστημα και να σταματήσουμε πλέον να βασιζόμαστε σε ειδικά ιδιωτικά εργαλεία ή την ε, ιδιωτική ε, επένδυση ε, γιατί οι ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επιλέξουν βάσει κριτηρίων απόδοσης και όχι βάσει κριτηρίων κοινής ωφελίας. Ε, επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να συνδυάσουμε τη συζήτηση με την ε, χρηματοδοτική και δημοσιονομική ικανότητα της ε, Ευρωζώνης, γιατί όλα αυτά τελικά αποτελούν δέσμοι. Όσον αφορά τώρα το τμήμα των δαπανών, εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογίες και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αλλά και να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό των επενδύσεων και λυπούμεθα γιατί ε, οι πόροι του, τα κονδύλια του ορίζοντα 2020 έχουν ε, μειωθεί. Αυτό είναι σφάλμα κατά την δική μας άποψη, γιατί πιστεύουμε ότι η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας προκύπτει από τα ε, επενδυτικά προγράμματα και τη χρηματοδότησή τους. Από την άλλη πλευρά δεν θα θέλαμε να εγκαταλείψουμε τον στόχο ενός παραγωγικού προγράμματος πλέον αηφόρου ε, και πλέον βιώσιμου ε, και να ε, βοηθηθούν αυτές οι νέες αρχές ενός νέου παραγωγικού συστήματος που θα βασίζεται ας πούμε σε εναλλακτικέ μορφές ενέργειας και όχι αυτά τα φαραωνικών διαστάσεων ε, προγράμματα τύπου ίτερ ή ε, ε, αγωγούς φυσικού αερίου ας πούμε που τελικά αφορά μια ενέργεια της οποίας η κατανάλωση μειώνεται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε συνάδελφε, κύριε Γκάγερ, τα τελευταία σας παρατηρήσεις ε, και ε, αν έχετε απαντήσει να δώσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η γνωμοδότηση πιστεύω πως ε, με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Γι' αυτό λοιπόν τη στηρίζω και συμφωνώ και με όλα τα σχόλια που άκουσα. Ως αναπληρωματικό μέλος αυτής της Επιτροπής να ξέρετε πως ε, είμαι πιο κοντά στα, ε, στις επιθυμίες σας και στις προσδοκίες σας από ό,τι τα άλλα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμού. Ε, ο κύριος Ρόιλ είχε δίκιο βέβαια. Κάθε επιτροπή έχει και το δικό της κατάλογο προτεραιοτήτων και μπορώ να καταλάβω αυτά που ζητάτε, όμως δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα έχουμε ένα δωράκι για την κάθε επιτροπή. Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω κάποιες υποσχέσεις και ανήκω στους πολιτικούς που ε, ξέρουν να λένε μόνο την αλήθεια. Πιστεύω πως ε, κύριε Ρόλη το πρόβλημα που έχουμε είναι το εξή. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομίε. Δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι τα κράτη-μέλη στην αρχή λένε ότι μεσοπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι πρέπει να τα βγάλει πέρα με λιγότερα λεφτά και ε, από το 2013 όμως και μετά με κάθε πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ακούγαμε ότι, ε, το αντίθετο. Ακούγαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι από τον προϋπολογισμό να τα βρούμε. Έχουμε δηλαδή περισσότερα έξοδα, λιγότερα έσοδα. Και έχουμε φτάσει, πιστεύω, σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό, λοιπόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν τι δεν θα χρηματοδοτούν από εδώ και στο εξή από τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό ή πρέπει να βρουν άλλους ε, τρόπους χρηματοδότηση διαφορετικά να ε, κάνουν περικοπές. Το Συμβούλιο έχει λάβει κάποιες αποφάσεις και φυσικά αυτές οι αποφάσεις πρέπει και να εφαρμοστούν, όμως ε, δεν μπορούμε να λέμε πως είμαστε σοβαροί πολιτικοί αν τα ρίχνουμε όλα στο Συμβούλιο. Ναι, θέλει να μετακαταστήσει ε, τόσους ε, πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν μπορούμε εμείς να διαθέσουμε τα κονδύλια κτλ. κτλ. Υπάρχουν προβλήματα από τον προπολογισμό. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το έργο μας, όμως πρέπει να είμαστε σοβαροί και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, μέχρι να φτάσουμε στο μη περαιτέρω, μπορούμε να προσπαθήσουμε, σίγουρα. Και χρειάζεται να είναι κάποιος καλλιτέχνης, έτσι, για να καταφέρει να ε, συνδυάσει όλες τις ε, προσδοκίες και ε, να καταφέρει να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει. Ναι, πρέπει να έχουμε και φαντασία για να το κάνουμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Τώρα, είτε. όσο και αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από αυτήν εδώ την Επιτροπή να είναι ε, λιγότερο, ε, να είναι περισσότερο συνετή μάλλον. Έχουμε πρόβλημα, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση και αυτό έχει οδηγήσει ε, να ακυρωθεί η απαλλαγή για αυτήν την υπηρεσία. Εάν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ΙΤΕΡ χρειάζεται λιγότερα κονδύλια για το 2017 από ό,τι είχαν εγκριθεί, ακριβώς διότι έχουν παραθυρηθεί αυτά τα προβλήματα, τότε τα μέσα, τα, τα κονδύλια τα οποία ε, έχουν δοθεί θα μειωθούν έτσι ώστε με αυτά να χρηματοδοτήσουμε κάτι άλλο. Δεν πρέπει να ε, νομίζετε ότι δεν πιστεύουμε αυτό το οικοδόμημα, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά ότι αντιθέτως θεωρούμε πως αυτά τα κονδύλια χρειάζονται πολύ ε, περισσότερο αλλού και θα χρησιμοποιηθούν με καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να ε, αμφισβητηθεί η ύπαρξη της ΣΥΤΑ. Τώρα, εάν η ίτερ στον επόμενο χρόνο λάβει λιγότερη χρηματοδότηση. Σίγουρα δεν είναι εύκολη αυτή η απόφαση, σίγουρα θα δυσαρεστήσει πολλούς, όμως θεωρώ πως σε καμία περίπτωση δεν ε, πρέπει να πιστεύουμε πως ε, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μας στην, στην Δεν πρέπει να έχουμε αυτή την άποψη. Τώρα, αγαπητέ συνάδελφε, μας είπατε για τα χρηματοδοτικά μέσα και ότι αυτά δεν είναι η λύση. Βέβαια, δεν είχαμε και παταγώδη αποτυχία. Υπήρχαν κάποια πράγματα που καταφέραμε να κάνουμε με χρηματοδοτικά μέσα. Κάτι καταφέραμε και εμείς να κάνουμε. Όμως, υπήρχε και μία προειδοποίηση Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε, διότι ισχύει για πολλά. Όταν χρησιμοποιούμε εναλλασσόμενα ταμεία, μπορεί αυτό να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως δεν πρέπει να γίνει ο κανόνας. Διότι, να ξέρετε, πως έχουμε και όρια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δεν γίνεται να λέμε άλλα στις Βρυξέλλες και άλλα στις πατρίδες μας. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες αλλού, δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδίους πόρους, για ε, ευθύνη κρατών μελών κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ να το μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στις εκλογικές σας περιφέρειες, τους ψηφοφόρους σας και να μην επαναλαμβάνετε ε, αυτό, το, αυτή την καραμέλα ότι ναι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσα λεφτά στις Βρυξέλλες αλλά εμείς δεν έχουμε κτλ. κτλ. Διότι αυτή ακριβώς η ρητορική μας οδήγησε εν μέρη σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητώ από σας περισσότερη ειλικρίνεια στο ε, τι περιμένουμε και τι κάνουμε με τα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι για τα σχόλια σας. Πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας. Και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια μας τα λέτε και σοβαρότητα είναι απόλυτα απαραίτητη αυτή η σχέση μεταξύ μας γιατί έτσι οικοδομείται η εμπιστοσύνη. Εκ των όνου κάνευ. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε από όσα μας λέτε και προηγουμένως και τώρα. Βεβαίω όλα τα σχόλιά σας τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ξέρουμε και ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες, αλλά και τα σημαντικότερα για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και πάλι, αγαπητέ συνάδελφε. Προχωρούμε τώρα λοιπόν στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη που είναι τα μέτρα κατοχήρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Είναι ένας νέος κανονισμός αυτός. Ο προηγούμενος ήταν το 2010. Δεν είχε λεφτείς εξ αρχής, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω δύο λόγια ως εισηγητής για το προφανές αυτό θέμα. Έχω το σχέδιο έκθεσής μου. Μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες πριν από λίγες μέρες και υπάρχει δηλαδή πλέον στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία εδώ κατά την αποψήμωσή του. Ξέρετε ότι είναι νομοθετικό αυτό το θέμα και έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τη γενική μας προσέγγιση ποια είναι. Αυτή που προτείνω εγώ τουλάχιστον. Ο νέος κανονισμός αυτός έχει τρία βασικά σημεία που είναι καινούρια, δεν υπήρχαν στον προηγούμενο. Αναφέρω λοιπόν τρία πράγματα μόνο, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Και οι δύο κανονισμοί, ιδιαίτερα ο τελευταίος, θα πρέπει κανονικά να βασίζονται σε λύσεις προσανατολισμένες στην αγορά. Αυτό είναι το σημαντικότερο για όλους μας. Δεν έχουμε αλλάξει τη βασική μας φιλοσοφία, ούτε, ούτε γνώμη. Αλλά στον προηγούμενο κανονισμό υπήρχε εθνική προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού κάθε κράτους μέλους. Στη συνθήκη Λισαβόνας και το, το άρθρο 194 ορίζει ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια ενεργειακού εμφοδιασμού των κρατών μελών είναι συναρμοδιότητα, συντρέχουσα αρμοδιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο και των κρατών μελών. Δηλαδή είναι κοινή αρμοδιότητα. Πρώτον, περιφέρειες. Εκεί νομίζω είναι το σωστό σημείο να κάνουμε ένα βήμα πρόοδο. Αν θέλουμε να σκεφτούμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο το εθνικό, για την ασφάλεια του εφοδιασμού μας με αέριο. Πρέπει να πάμε προς την κατεύθυνση αυτή, να σκεφτούμε και τις περιφέρειες και τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πλήρη αρμονία με τη συνθήκη. Για να μεγιστοποιήσουμε όμως τα ευεργετήματα για τις περιφέρειες, για τη συνεργασία, και να έχουμε και ευελιξία στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προσέθεσα την έννοια του διαδρόμου για τον επίγοντα εφοδιασμό. Σε συνεργασία με το ENSO G, που είναι ε, οι ε, διαχειριστές των δικτύων ε, μεταφοράς. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε τους διαδρόμους αυτούς και να τους εντοπίσουμε και να επιτρέψουμε τη συνεργασία διαφόρων διαδρόμων που μπορεί να είναι λίγα, λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να φτιάχνουμε νέους αγωγούς. Καμιά φορά αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε ε, νέες διασυνδέσεις διασυνοριακές ο κανόνας είναι να εντοπίσουμε τους υφισταμένους διαδρόμους και διάβλους και να υπάρχει δυνατότητα επίγουσας συνεργασίας όπου θα συνεργάζονται τα κράτη-μέλη, ένα-δύο που βρίσκονται στη διαδρομή του αγωγού και αν συνεργαστούν θα μετριαστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από μια μεγάλη κρίση στην παροχή φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί μιλώ για μεγάλη κρίση, διότι μίζωνα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να λύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις δύσκολες καταστάσεις ε, με τη συνεργασία της δικής μας αγοράς, έτσι, μίζωνες ε, κρίσεις. Πολύ σημαντικό. Δεύτερο θέμα, η αλληλεγγύη. Κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί για να ε, καταστεί πιο ισχυρή και ανθεκτική όταν υπάρχουν ε, προβλήματα στις τιμές. Αλλά όταν υπάρχει κρίση να χρησιμοποιείται αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης ως έσχατη καταφυγή. Τι σημαίνει αυτό. Ε, η αλληλεγγύη σταματάει να είναι αξία απλώς και θεωρητική και γίνεται νομικός ε, μηχανισμός. Και βέβαια προτείνω εναρμονισμένο ε, ορισμό για να καλύπτεται ε, ένας μικρός αριθμός τελικών καταναλωτών και χρηστών. Το ίδιο ισχύει για τα κράτη-μέλη. Δεν μιλάμε για τους ίδιους αριθμούς, αλλά για το ίδιο είδος χρηστών. Προτείνω ένα ορισμό δηλαδή για τον τελικό καταναλωτή για πολύ μικρές ε, κατηγορίες. Επαναλαμβάνω όχι σε απόλυτους αριθμούς. Και το τρίτο βεβαίως είναι η διαφάνεια και συνδέεται απολύτως και πάρα πολύ στενά με κάτι που ονομάζουμε πλήρη ε, συμφωνία όλων των συμβάσεων με το κείμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται κοινοποίηση σε κρίσιμες περιπτώσεις εμπορικών συμβάσεων και συμβολέων που πρόκειται να υπογράψουμε με προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Uh, Περί αυτού πρόκειται, δεν μιλάμε για τον ιστορικό αφοδιασμό, μιλάμε για τρίτους προμηθευτές. Έτσι το ορίζω λοιπόν και έτσι είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και προτείνω να αντικατασταθεί το 40% της κατανάλωσης από 40% εισαγωγών και να αποκλείονται χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ΕΟΧ, ε, από το χαρακτηρισμό τους ως εξωτερική εταίρη. Δεν είναι εξωτερική, εσωτερική είναι ο ε, ΕΟΧ τώρα. Δεν μιλάμε για αυτές τις χώρες. Γιατί διέπουν ακριβώς τους ίδιους, ίδιοι κανόνες ε, τον ΕΟΧ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τρίτες χώρες αυτές με την έννοια αυτή. Λοιπόν, αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνω σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ακούμε τους σκιώδες τώρα. Η κυρία Γκρίφιν από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγήτα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούζεκ για την εργασία του. Πιστεύουμε ότι το θέμα της βιωσιμότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί και βεβαίως και το θέμα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι σημαντικό έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις εξαγωγές φυσικού, ε, εισαγωγές διορθώνω φυσικού αερίου. Οπωσδήποτε θα πρέπει να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη και οι στόχοι του κλίματος και οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να μειωθεί η κατανάλωση αερίου. Θα πρέπει επίσης να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ε, ανάγκες ε, κατανάλωσης φυσικού αερίου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, ανάμεσα στο φυσικό αέριο και την, την ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος, η προσέγγιση του εισηγητή για την περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σωστή. Τα περιφερειακά προγράμματα δεν θα ε, πάρουν τη θέση, δεν θα αντικαταστήσουν ε, τα εθνικά προγράμματα. Ωστόσο, η διαμεθοριακή συνεργασία μπορεί να είναι σωτήρια σε περίπτωση ε, ιδιαίτερων καταστάσεων και διακοπής της παροχής ναι, και ε, ε, επομένως σε αυτή την περίπτωση η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, δεν θα πρέπει να εμποδιστεί μεγαλύτερη και εντονότερη συνεργασία έτσι, μεταξύ των χώρων έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού. Είναι σημαντικό οι ε, περιφέρειες οι οποίες θα έχουν δημιουργηθεί ε, να μην αποτρέπουν οποιασδήποτε άλλες συνεργασίες μεταξύ χωρών που δεν συμμετέχουν στην ίδια ε, περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Τζέζακ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητά που παρουσιάσατε αυτό το σχέδιο έκθεσης το οποίο όπως όλοι διαπιστώνουμε είναι πολύ καλό και ε, ε, λεπτομερές. Θα σας πω την άποψή μου τώρα όσον αφορά το προσχέδιο αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κύριος στόχος ε, της προσπάθειας θα είναι να μειώσουμε την ευαισθησία μας και την εξάρτησή μας από την εξωτερική ε, προμήθεια και επίσης ε, να προστατεύσουμε τους προστατευόμενους ε, πελάτες και να δημιουργήσουμε την αλληλεγγύη αυτή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και διαφάνεια για όλες τις συμβάσεις με ξένους πάροχους. Συμφωνώ την γραμμή που, με τη γραμμή που έχει πάρει ε, ο ε, εισηγητής μας και όσον αφορά την περιφερειοποίηση και όσον αφορά την ρήτρα αλληλεγγύης. Ε, ε, τα stress τεστ της Κομισιόν έχουν ε, δείξει ότι ορισμένες περιφέρειες δεν έχουν την ανθεκτικότητα την οποία θα έπρεπε να έχουν και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα και τις δυνατότητες. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία εν λεπτομερία. Συμφωνώ ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τούτη τη στιγμή δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, ε, ε, ε, δημιουργηθεί ένας, καλύτερης, ένας μηχανισμός μεγαλύτερης συνεργασίας. Ε, επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφέρειες οι οποίες θα έχουν προληπτικά προγράμματα καθώς επίσης και προγράμματα σταθερότητας. Όσον αφορά τώρα τις ε, ε, καταστάσεις έκτακτης ε, ανάγκης, εδώ θα πρέπει να εισαχθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ρήτρα αλληλεγγύης στον κανονισμό αυτό, γιατί πιστεύω ότι ε, αυτή η αρμοδιότητα είναι κοινή και θα πρέπει να βασίζεται ε, στον κανόνα της ε, συνεργασίας. Χαίρομαι γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την διαφάνεια των συμφωνιών και των συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν αυτές οι συμφωνίες. Πιστεύω ότι οι συμβάσεις και οι συμφωνίες, αυτές που υπογράφονται δηλαδή με παρόχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ε, ε, είναι διαφανής έτσι ώστε να μπορούν όλοι να τις ελέγξουν. Βεβαίως θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες οι οποίες στόχο θα έχουν την περαιτέρω ενδυνάμωση της ασφάλειας εφοδιασμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εξ ονόματος κυρίου Τσαλίξκα θα ήθελα ε, να υπογραμμίσω ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα της ε, ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για έκτακτες εξαιρετικές καταστάσεις που στατιστικά μπορεί να συμβούν μία φορά τη δεκαετία. Αναφερόμαστε ε, σε ε, διαχείριση κρίσης και όχι σε συνηθισμένες ε, διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί η ρήτρα αλληλεγγύης έτσι ώστε ε, να ε, συνεχίσει η παροχή ενέργειας ε, στις πιο ευαίσθητες ομάδες, στις πιο ευαίσθητες βιομηχανίες και στα νοικοκυριά. Αλλά ακόμα και αν μιλάμε για αντιμετώπιση κρίσης θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να έχουμε προσέγγιση τύπου αγοράς. Ναι, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβλέψουμε και κάποια ορθή ή αποζημίωση, γιατί αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Ε, το, ε, η διάνοιξη ε, οδών διεμπορίας είναι κάτι σημαντικό και οι στρατηγικές υποδομές επίσης είναι κάτι που ο εισηγητή, ο Σκιώδης από την πολιτική μας ομάδα θεωρεί κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάβο ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Τούρμες Ευχαριστώ Πρόεδρε, εξ ονόματος του κυρίου Τούρμες, ε, να πω ότι ζητά συγγνώμη γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να ε, ε, παρίσταται στη συζήτηση. Πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά ενέργειας και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού είναι καλή πρόταση ο νέος κανονισμός ε, θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη βάσει των ε, περιφερειακών συνεργασιών ε, εμείς συμφωνούμε με την προσέγγιση της Κομισιόν όσον αφορά ε, την ε, περιφερειακή συνεργασία. Ε, είναι σημαντικό να πούμε ότι το γεωγραφικό εύρος της περιφερειακής συνεργασίας είναι προκαθορισμένο έτσι ώστε να μπορούν να καθοριστούν προγράμματα δράσης και, και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουλέψουν βάσει κοινών σεναρίων όσον αφορά περίπτωση ε, ε, διακοπής του εφοδιασμού. Στον κανονισμό θα πρέπει να βρεθεί ένας ισχυρός μηχανισμός βάσει του οποίου θα λειτουργεί σωστά η αρχή της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι προστατευμένοι πελάτες που κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι τα νοικοκυριά ε, και ορισμένοι ε, ε, αστικοί και μη αστικοί πελάτες που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καθώς επίσης και ορισμένες υπηρεσίες κοινή ωφελία. Ο ορισμός λοιπόν του προστατευόμενου και μη θα πρέπει να είναι σαφής. Ε, σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να επαναπροωθείται το αέριο προς γειτονική χώρα των οποίων οι προστατευόμενοι, τις οποίες οι προστατευόμενοι πελάτες έχουν υποστεί διακοπή της ροής αερίου. Όμως το κείμενο δεν αναφέρει ε, την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα και ε, την ενεργειακή απόδοση, συγγνώμη, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει κάτι τέτοιο να αναφερθεί. Ο κανονισμός επίσης λαμβάνει υπόψη την φθήνουσα πορεία της ζήτησης του φυσικού αερίου και λαμβάνει υπόψη και τα, όλα τα μέτρα τα εθνικά και τα προγράμματα τα εθνικά όσον αφορά ε, την μείωση της εξάρτησης ε, από τις ε, εισαγωγές. Πιστεύουμε ότι τα δύο αυτά στοιχεία θα πρέπει καλύτερα να αναφερθούν στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλάγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι, εμείς δεν συμφωνούμε και πάρα πολύ ε, για να μην πω καθόλου με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αέριο, το φυσικό αέριο και ο εισηγητής προς την ίδια κατεύθυνση είναι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να έχει θετικά στοιχεία, αλλά συνολικά δεν συμφωνούμε με την έκθεση. Πάντως ευχαριστούμε τον εισηγητή για την προθυμία του να ανταλλάξουμε απόψεις και ήταν πάρα πολύ θετική συνεργασία μας. Ε, έλεγα ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στα εξής. Αφενός και σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες αγοράς για να ρυθμίζονται έκτακτες καταστάσεις που από τη φύση τους είναι ε, διαφορετικές και δεν θα μπορεί να τις διαχειρίζεται η αγορά που είναι τόσο ε, ασταθής. Επίσης ε, όταν ε, αυξάνονται η αγωγή φυσικού αερίου και η χρήση φυσικού αερίου και κατανάλωση, αυξάνεται και η εκπομπή ε, διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια και τη διαφορά από περιφέρεια σε περιφέρεια, μπορεί να χαρακτηριστούν ορισμένοι αγωγοί φυσικού αερίου στρατηγικές υποδομές και τελικά να καταλήξουμε σε μια κατάσταση εμπλοκής όπου θα είμαστε δεμένοι χειροπόδερα ε, με αυτή τη μορφή ορυκτού καυσίμου. Αν θέλουμε να εισαγάγουμε την αρχή της αλληλεγγύης, αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά θα πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα και ε, στην ενεργειακή πολιτική να το δούμε συνολικά ε, στην Ευρώπη και όχι μόνο όταν ε, σφίγγουν τα πράγματα και είναι κρίσιμα. Ε, οι προστατευόμενοι πελάτες είναι κάτι καλό. Να υπάρξει ευρωπαϊκός ορισμός όπως προτείνει ο εισηγητής, χωρίς αποκλεισμούς όμως για να προστατεύονται περισσότερο οι πολίτες που έχουν περισσότερη ανάγκη για τις βασικές ανάγκες προς όφελος όλης της κοινωνίας. Και τελειώνω. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι θεωρούμε εκ των όνων στο κείμενο αυτό να συμπεριληφθούν μέτρα μείωσης της κατανάλωσης και άρα και μείωσης της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ενδιαφέρουσες εκεί συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάπελη, αυτό λέγω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα τρία κύρια σημεία που βλέπουμε διαφορές έχουν ήδη αναφερθεί. Αλληλεγγύη, διαφάνεια. Υπάρχει και η πρόταση για τον ορισμό των, ε, κριτήριο, των κριτηρίων για τις ε, διάφορες περιφέρειες. Ε, εδώ Έχω τις αμφιβολίες μου. Είπα ότι πρέπει να ε, συσταθεί μια περιφέρεια νοτιοδυτικής Ευρώπης η οποία καλύπτει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ένωση και από την άλλη ένας άξονας βορρά-νότου που, φτάνει, που αρχίζει από την Ουγγαρία και φτάνει ε, στη Σλοβενία. Δεν νομίζω πως αυτό θα μας οδηγήσει στον στόχο μας. Εδώ πιστεύω αντίθετα πως χρειαζόμαστε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, bottom-up, έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Αυτή η πρόταση που έγινε για, τα, για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τους διαδρόμους έκτακτης ανάγκης, θεωρώ πως είναι καλή. Αλλά ο ορισμός των περιφερειών έτσι όπως βρίσκεται στο κείμενο ε, μου φαίνεται πως χρειάζεται βελτίωση, πως είναι αναγκαίο μάλιστα να βελτιωθεί έτσι ώστε να... Ε, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σίγουρα χρειάζεται βελτίωση στις υποδομές, λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ρήτρα αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη μας είπατε ότι είναι ένα μέτρο ε, τελευταίας λύσης. Χρειάζεται όμως να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ορίζουμε αυτήν την ρήτρα αλληλεγγύης, αλλά και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείται και να ε, διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται ορισμένα πρότυπα ε, ασφαλείας. Διαφορετικά ε, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Είναι, πιστεύω, αυτό πολύ σημαντικό τώρα στην υποβολή εκθέσεων στα πλαίσια του REMIT. Χρειάζεται, πιστεύω, να αναφερθούν στοιχεία όπως η ελάχιστο, ο ελάχιστος όγκος παράδοσης, προθεσμίες, όροι της ε, σύμφασης κτλ. Αυτά δεν έχουν αναφερθεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν έναν μεγάλο ρόλο και εδώ υπάρχει και αντίστοιχη οδηγία για τις ε, υποδομές. Έτσι όπως έχει η πρόταση, δεν γίνεται ο πάροχος να είναι επίσης υπεύθυνο και για τις υποδομές. Αυτό σίγουρα δεν θα μας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν θα μας οδηγήσει σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε, αλλά πρέπει ε, αντιθέτως να βρούμε λύση έτσι ώστε η δικτύωση μεταξύ κρατών μελών να ε, πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγια. Κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η εργασία του Πρόεδρου μας ε, για ένα τόσο σημαντικό και στρατηγική σημασία θέμα, ε, η εργασία που έκανε, λέω, ο Πρόεδρος, όπως και η συνάδελφος Τερέζα Γκρίφτη είναι πραγματικά ε, εξαιρετική, έτσι ώστε να εξευρεθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση. Θα ήθελα λοιπόν να αξιολογήσω θετικά την εργασία αυτή γιατί ε, πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός, ε, ιδίω ε, όπως ο Σάβελα Κουάδρας και άλλοι που δούλεψαν για τον προηγούμενο κανονισμό ξέρουν πολύ καλά πώς, πόσο δύσκολο είναι κάποιες γενικές αρχές να συγκεκριμενοποιηθούν σε μηχανισμούς και μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της αλληλεγγύης που πλέον γίνεται νόμος μια υποχρέωση λοιπόν νομική βάσει συγκεκριμένων ε, και σαφώς καθορισμένων ε, διαδικασιών. Επίσης ο ορισμός των προστατευόμενων ε, ή προτιμησιακών πελατών. Ε, αυτές ε, είναι, αυτοί είναι ορισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Υπάρχουν όμως δύο σημεία δύο σημεία λέω τα οποία δεν με ικανοποιούν απολύτως ε, και εδώ θα πρέπει μέσω των τροπολογιών να ε, τροποποιήσουμε λίγο την κατάσταση. Θα πρέπει να βρούμε την συμφωνία ανάμεσα στα εθνικά προληπτικά προγράμματα και τα περιφερειακά. Ε, να δούμε ποια, ποιες είναι οι δράσεις οι οποίες θα αφορούν την περιφερειακή συνεργασία ε, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, χωρίς όμως ε, να διακόψουμε, να διαγράψουμε οποιαδήποτε σχέση ε, με τα εθνικά προγράμματα. Η διασύνδεση θα πρέπει να είναι όσο γίνεται σαφέστερη και πιο συγκεκριμένη. Δεύτερον, ε, το θέμα, αυτή η ιδέα των περιφερειακών ε, ενώσεων αυτών των περιφερειών, λοιπόν, εγώ το βλέπω και από πλευράς της χώρας μου, αλλά όχι μόνο νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να ε, παραμείνουμε σε μια άκαμπτη γεωγραφική ε, συνεργασία όταν μιλάμε για αλληλεγγύη γιατί ε, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές αρχές και αυτό ακούστηκε και από την Τερέζα δηλαδή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία με όμορες περιοχές ναι αλλά υπάρχουν και χώρες οι οποίες ε, ε, έχουν σύνορα με τρίτη χώρα πριν ε, φτάσουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ας πούμε σκέφτομαι την Ελβετία. Επίσης υπάρχουν χώρες με τις οποίες έχουμε ήδη διασυνδέσεις που περνάνε μέσα από τρίτη χώρα. Και επίσης ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το παρόν ε, σύστημα των ε, δικτύων. Δεν ξέρω εάν, κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό των διαδρόμων για τις έκτακτες επίγουσες καταστάσεις. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ με την έκθεση με ορισμένες διορθώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και πρόεδρο μας. Πραγματικά είναι πολύ καλή η έκθεση. Γίνεται λόγο για νέα εργαλεία και για νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας που εργάζονται εδώ και χρόνια για τα θέματα αυτά ε, γνωρίζουν πως έχει κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ ευτυχής. Ε, ε, ωραία είναι η περιφερειακή συνεργασία, αλλά αν μιλάμε πρώτα για την αγορά και στην πραγματική ζωή αναφερόμαστε στις αγορές, η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό μας είναι το κέρδος. Άρα η συνεργασία μεταξύ περιφερειών, η ελεγγύη είναι ωραία λόγια, αλλά ε, οι αγορές την κερδοφορία επιζητούν και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να παρακάμψουν ορισμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένες επιθυμίες. Όλα αυτά είναι επόμενα και φυσιολογικά. Ε, δεν μιλάμε μόνο για τις υποδομές αλλά και για την ανταγωνιστικότητα κάθε κράτους μέλους. Εάν ε, μειωθεί η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους μέλους ε, στο βωμό της αλληλεγγύης, το κράτος χάνει έσοδα. Οπότε οι πολίτες δεν θα χαρούν ιδιαίτερα αν μάθουν ότι για λόγους χ αλληλεγγύης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ψ χρειάστηκε να υποστηρίξουμε ένα γειτονικό κράτος και να χάσουμε εμείς πόρους από τον προϋπολογισμό μας. Θα πρέπει να συζητήσουμε τελικά ποιος θα φέρει την ευθύνη όλων αυτών εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για την ε, δημιουργία της αγοράς ενέργειας και ειδού πώς έχει τώρα η κατάσταση χτίσαμε ένα τερματικό σταθμό για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και έπεσε τιμή του αερίου. Τώρα εμείς τι να το κάνουμε αυτό. Χαίρομαι πολύ για την Ελβετία που είναι στο κέντρο της Ευρώπης και μπορεί να ε, εποφελείται ε, και να εκμεταλλεύεται τις υποδομές των γύρω-γύρω χωρών, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν άλλη γεωγραφική θέση και δεν απολαμβάνουν αυτή τη δυνατότητα. Για να εξασφαλίσουμε ε, τον εφοδιασμό θα πρέπει να είναι αρμόδια και υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας υποστηρίζω σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι φορά τώρα το φυσικό αέριο, αυτό καθ' αυτό, πριν από λίγες εβδομάδες στην Επιτροπή μας μας απασχόλησε το θέμα, ιδιαίτερα ε, ε, αυτά που λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Για τις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Αν φτιάξουμε νέους αγωγούς φυσικού αερίου, θα εξαρτηθούμε από άλλο προμηθευτή. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ανεξάρτητοι. Και η εξάρτηση αυτή θα έχει ορίζοντα 40 ετών, 50 και παραπάνω. Το θέμα του φυσικού αερίου είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει από κοινού με τον εφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί σε περίπτωση κρίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσανατολίσουμε τη βιομηχανία μας προς ε, συγκεκριμένες αποφάσεις. Όταν υπάρχει κρίση στο φυσικό αέριο, να χρησιμοποιούμε το ρεύμα, το ηλεκτρικό που θα είναι πιο φτηνό ή θα έχει περισσότερο. Έτσι θα αυξήσουμε και την ανεξαρτησία μας και την ασφάλειά μας για τον εφοδιασμό σε ενέργεια, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Υποστηρίζω την έκθεσή σας κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλύτερη από την αρχική πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκιούρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν, κυρίως τον εισηγητή και να τον συγχαρώ μάλιστα. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι ύψης της σημασίας και αρκετοί από εμάς από το 2006, από την πρώτη δηλαδή κρίση του φυσικού αερίου ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και ακριβώς σκεπτόμενοι την κρίση αυτή θα πρέπει ε, να θεωρούμε τον ε, νέο κανονισμό, τη νέα ρύθμιση, όχι ως ε, φορτίο, αλλά ως μια λύση για το πρόβλημα. Πρέπει να στηρίξουμε την συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έτσι διαβάζω και συμφωνώ. Όμως τα κράτη-μέλη και όμως τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει ε, να ε, ρυθμίσουν το πώς ε, θα το κάνουν αυτό. Χρειάζεται όμως και αρκετή ευελιξία, ιδιαίτερα όσον αφορά την διασυνοριακή συνεργασία. τώρα, η ρήτρα αλληλεγγύης. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ένα κράτος μέλος δηλαδή να την θέτει σε ισχύ μόνο όταν έχει εξαντλήσει τους δικούς του ενεργειακούς πόρους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη ρήτρα αλληλεγγύης. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε η κατανομή του ε, βάρους να είναι ίση σε όλους και όχι να έρθουν κράτη-μέλη σε ε, δύσκολη θέση και μιλώ για τα κράτη-μέλη τα οποία ε, γεωγραφικά βρίσκονται σε τέτοιες νευραλγικές επλέσεις ή δεν έχουν ένα ε, σύστημα αντιμετώπισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφαν Μόζερ τώρα θα μας μιλήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην συζήτηση για τον κανονισμό για το φυσικό αέριο. Όπως και αρκετά ε, μέλη, έτσι και εμείς θεωρούμε τον κανονισμό αυτό ως ένα κομμάτι της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτό μαζί με τα μέτρα για το περιβάλλον, με την ενεργειακή απόδοση και ένα μέρος της στρατηγικής για το 2020 και 2030. Ένα ε, αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας είναι η ενεργειακή απόδοση και ο η ασφάλεια του φωδιασμού με φυσικό αέριο. Μάλιστα θα έλεγα πως ε, εκεί βασίζεται και όλη η πρόταση. Έπειτα, πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η εσωτερική αγορά. Είναι το, το κύριο μέσο για να επιτεύξουμε τους ε, στόχους μας και χρειάζεται να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως ε, όλο το περιεχόμενο του, της δέσμης μέτρων. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μπούζεκ, μέχρι τώρα έχουμε δει ότι τα κράτη-μέλη οθέτησαν μία ε, εθνική προσέγγιση. Χρειάζεται όμως περιφερειακή προσέγγιση. Χρειάζονται όχι μόνο εθνικά μέτρα, αλλά περιφερειακά. Ε, χρειάζεται ανάλυση, αλλά όχι μόνο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και πολύ καλό είναι να υπάρχει μια ανάλυση εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορούμε να ε, δούμε ποιους ε, διαδρόμους έκτακτης ανάγκης θα μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά πιστεύω πως αυτό είναι συμπληρωματικό και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την κύρια την κύρια πρόταση, η οποία είναι η περιφερική συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν και ως συμπληρωματικό μέτρο, ναι, το καλωσορίζω. Τώρα, συμπληρωματικότητα, πιστεύω πως εδώ είναι το σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και ο καθένας να χρησιμοποιεί τα δικά του ε, πλεονεκτήματα. Έτσι πρέπει να είναι μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ε, μην δράσουμε καθόλου, διότι οι συνέργειες έτσι δεν θα υφίσταται πλέον. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχει έρθει η ώρα σε αυτήν εδώ την ε, νομοθετική περίοδο να αποφασίσουν και να αναλάβουν δράση. Δεν χρειάζεται να αναβάλουμε τις αποφάσεις, αλλά πρέπει να γίνει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουν τώρα ποιο είναι ένα κατάλληλο ε, νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά, εάν αναβληθούν οι αποφάσεις, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα πολλά. Θα περάσουν χρόνια συζητήσεων μέχρι να αποφασίσουμε ποιος είναι αρμόδιος, ποιος πρέπει να κάνει τι. Αυτό εμείς θεωρούμε πως είναι αναποτελεσματικό. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε η πρότασή μας να συνοδεύεται από αξιολογήσεις ομοτήμων και από διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, με τα κρατημέλη, με τον ε, ε, κλάδο της βιομηχανίας, με την ενεργοβόρο βιομηχανία, έτσι ώστε να αποκομίσουμε μια ε, σωστή και πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ανάγκες και να φροντίσουμε να μην ε, υποστεί Ζημιά η έννοια αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Πολλές φορές οι ε, ενδιαφερόμενοι φορείς μας λένε ότι θέλουν να καταλάβουν και να ξέρουν τι θα γίνει και δεν θέλουν να βρεθούν ε, πρωτοτελεσμένου γεγονότος και προεκπλήξεων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η αναβολή είναι λάθος. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα απλά αφήνοντας τα κατά μέρος. Τώρα, όπως είπε και ο Μπούζεκ, το καινοτόμο στοιχείο εδώ είναι ότι ε, περνάμε από τα λόγια στις πράξεις. Και η ρήτρα αλληλεγγύης είναι κάτι καινούργιο, αλλά όπως είπατε κι εσείς είναι μια λύση της ε, είναι μια τελευταία λύση. Πρέπει να προβλεφθεί κάποια αποζημίωση, κάποια συμπληρωματικά μέτρα. Γι' αυτό χρειάζονται και άλλες ε, συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε όσες πληροφορίες χρειαστούμε. Χρειάζεται ένα εναρμονισμένο πλαίσιο επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται διαφάνεια όσο για τη διαφάνεια. Πιστεύω ότι στην πρότασή μας προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία, να εντοπίσουμε σε εκτιμήσεις ε, κινδύνου, τους ε, κινδύνους και να προσπαθήσουμε να τους ε, αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Γι' αυτό προσπαθήσαμε στην πρότασή μας να τηρήσουμε τα πρότυπα του ΠΟΕ και να απαγορεύσουμε τις διακρίσεις εις βάρος εταιριών από έξω εντός. Αυτό δηλαδή είναι μια προσπάθεια για να ε, αποφευθεί η ανασφάλεια, νομική ανασφάλεια, έπειτα. Είναι διπλής κατεύθυνσης η πρόταση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ε, τα κράτη και από τα κράτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή, αυτός ο αμφίδρομος χαρακτήρας διασφαλίζει, πιστεύω, την, ε, τον ενεργειακό εφοδιασμό με αέριο. Τώρα, όσο για τη σύνδεση αερίου με ηλεκτρισμό. Εδώ χρειάζεται να προβλέψουμε την επαρκή προστασία των ε, ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είστε σίγουροι πώς συμπεριλαμβάνετε στην πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ όλους, σκιώδες ηγητές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προφανές ότι η συμφωνία από ε, όπως όλες αυτού του είδους οι συμφωνίες είναι απολύτως απαραίτητες. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική ε, υποστήριξη για αυτό το σχέδιο Έκθεση, Βεβαίως ε, περιμένω και ε, πολλέ τροπολογίε, ε, όπως πάντα. Αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα λόγια που μου είπατε. θα κάνω και κάποιες προσθήκες βέβαια, τώρα δεν μπορώ να τις αναφέρω όλες. Κυρία Γκρίφιν, βεβαίως μικρότερη εξάρτηση αυτό είναι κάτι προφανές ε, που θα οδηγήσει βέβαια σε λιγότερες ε, ε, εισαγωγές, τουλάχιστον στις περιπτώσεις της αλληλεγγύης. Αυτό θα πρέπει να διαλευκανθεί, όπως και το σύστημα της των διαδρόμων για τις έκτατες ανάγκες τώρα. Τώρα όσον αφορά αυτά που είπε η Κομισιόν, ε, εγώ κατέδειξα κάποια στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά ε, για την προσέγγιση της ε, αγοράς. Κύριε Γιάβολ, οι αποζημιώσεις. Εξ ονόματος του κύριου Τούρμες θα είπατε αυτά. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν ακόμα οριστεί αυτά σαφώς και χρειάζομαι τη στήριξή σας. Γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Και ο κύριος Μπαλσίτης αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα, το θέμα ε, της αποζημίωσης σε περίπτωση ε, αλληλεγγύης ε, θα είναι βεβαίως σε περίπτωση ε, ιδιαίτερου προβλήματος και σαν ίστατη προσφυγή και ευελπιστώ ότι δεν θα, δεν θα χρειαστεί ποτέ να προσφύγουμε σε αυτή την λύση και σε αυτούς τους διαδρόμους για τις επίγουσες καταστάσεις αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και είναι απολύτως απαραίτητη και αποζημίωση. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε και από τον κύριο Μπενιτόπουλο και από την κυρία κυρία Κάπελ και από τον κύριο Γιούρκα και από την κυρία Τόια και ίσως και από κάποιον άλλον. Το θέμα των περιφερειών. Πρέπει να σας πω, στις συζητήσεις που κάνουμε με τους και συγητές ή μεταξύ μας, μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν ως έχει. και να σκεφτούμε λίγο ε, ε, τις ομάδες χωρών αναπεριφέρεια και να μην ε, σκεφτούμε μόνο με όρους ε, εθνικής προσέγγισης που είναι βεβαίως κάτι δυνατό, κάτι μπορεί να γίνει. Βεβαίως όλες αυτές οι περιφέρειες είναι ανοιχτέ στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν ε, περιφέρειες γιατί όπως ε, είπε και η Κομισιόν είναι δύσκολο να περάσουμε από το επίπεδο ε, του κράτους μέλους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως μας μένει η περιφερειακή προσέγγιση και είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτό το σκεπτικό. Εάν προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα εθνικά προγράμματα, αυτό θα είναι κάτι πολύ δύσκολο, α, τουλάχιστον στα σημεία κίνηση Να ξεκινήσουμε λοιπόν διαφορετικά. Το ίδιο συμβαίνει και με εμά, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμεί είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερχόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Κάθε ένα από εμά έχει μία πρόταση η οποία προέρχεται από τη δική του κυβέρνηση, από τη δικιά του ε, χώρα μέλος, από τη δικιά του μόνιμη αντιπροσωπεία. Γνωρίζουμε τις προτάσεις, ε, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις, ε, γιατί εάν πάρουμε ο καθένας από τις κυβερνήσεις του και τις μόνιμες αντιπροσωπείες 28 προτάσεις, τότε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Είναι αδύνατο να βρούμε συμφωνία. Επομένως εδώ έχουμε μία πρόταση για να αλλάξουμε την προσέγγιση μας. Εγώ ε, δεν έχω τίποτα εναντίον το, της ε, εθνικής προσέγγισης, αλλά τα κράτη-μέλη, ε, οι χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να σκεφτούν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή όχι να βάλουν τη μία δίπλα στην άλλη ή να συνδυάσουν 5 και 6 και 7 διαφορετικά προγράμματα, γιατί αυτό δεν θα κάνει μία καλή προσέγγιση. Ε, τα συστήματα, οι διαχειριστές ε, των ε, συστημάτων μεταφοράς βεβαίως είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν. Επομένως, περιμένουμε προτάσεις από τις περιφέρειες έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε πιο συνεχτικές λύσεις. Η φυσική, ας πούμε, προσέγγιση ε, είναι πολύ πιο προχωρημένη στον τομέα της ε, ε, ή του ηλεκτρικού είναι αυτή η προσέγγιση bottom-up που ανέφερε η κυρία Κάπελ. Αλλά στο, στην περίπτωση φυσικού αερίου δεν είναι τόσο εύκολο να ακολουθήσουμε την ίδια οδό. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε, να στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Η αλληλεγγύη, οι προστατευόμενοι πελάτες, η διαφάνεια, όλα αυτά τα αναφέρατε. Πολύ δουλειά μένει, πολλή συζήτηση έχουμε ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Πολύ δουλειά όπως έλεγα μας μένει, θα ανασκουμποθούμε και ε, θα ε, ε, προχωρήσουμε. Στη Σλοβακική Προεδρία, μάλλον η Σλοβακική Προεδρία, ε, ε, μπορώ να σας το πω από τώρα, είναι έτοιμη για πολύ σκληρή δουλειά και αυτό περιμένουμε και σε αυτό προσδοκούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. 15 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ε. Αύριο, τι μου λέτε, λέει ο πρόεδρος. Αύριο λοιπόν, για φαντάσου, πω πω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει λέει ο Πρόεδρος, 15 Ιουνίου 12 το μεσημέρι λοιπόν λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Έχουμε τώρα το επόμενο θέμα, είναι ο κύριος Αντράζο Γκιούρκ στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου είναι θέμα σχετικό με τον ε, κανονισμό για τις έκτακτες ε, ε, περιπτώσεις φυσικού αερίου, κανονισμός SOS. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου για τα σχόλια και τι προτάσει που κάνατε. Πιστεύω ήταν πολύ σημαντικό να διαβάσω όλα σα τα σχόλια πρωτού ολοκληρώσω την ε, έκθεση. Ε, καταρχάς θα αρχίσω με ένα σχόλιο για, τη σχόλιο για τη μεθοδολογία. Επικεντρώθηκα μόνο στην ε, ενέργεια και στην αποθήκευση φυσικού αερίου. Γι' αυτό λοιπόν και περιορίστηκα και δεν ανέφερα όλα τα πράγματα τα οποία αναφέρατε εσείς. Ε, φυσικά διότι υπάρχει και ένας περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος ε, μιας έκθεσης. Αυτή η έκθεση στηρίζεται στην ε, έκθεση για την Ενεργειακή Ένωση, την ΜΑΜΑ έκθεση και εκεί ήμουν σκιώδης εισηγητής και θυμάμαι πολύ καλά τις έντονες διαβουλεύσεις που ε, είχαμε κάνει και σίγουρα δεν θα ήθελα να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω ότι στο σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνονται αρκετές προτάσεις. Έχω κάνει μία εξαίρεση όμως και αυτή αφορά τον αγωγό North Stream. Υπήρξαν ορισμένα προκλητικά σχόλια. Ε, ενήργησα με τον τρόπο που ενήργησα διότι προσπάθησα να έρθω σε έναν ε, συμβιβασμό με τους κοιόδης εισηγητές καλύτερα τώρα παρά αργότερα. Τώρα, επί της ουσίας, σε γενικές γραμμές το σχέδιο έκθεσης στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επικροτεί τις προτεραιότητες. Καταρχάς, τη συμπλήρωση των ελλείψεων στις υποδομές, προώθηση του διεθνούς εμπορίου ενέργειας, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος επέκτης και το υγροποιημένο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως ενεργειακή πηγή. Στηρίχτηκα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχος μου ήταν να ενισχύσω το μήνυμά της και να τονίσω κάποιες ε, συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας ε, της μείωσης στην εγχώρια παραγωγή. Σε ορισμένα κρατημέλη η εξάρτηση στο φυσικό αέριο φτάνει το 100% με ε, καμία πολλές φορές εναλλακτική λύση με ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις. Τα ε, πιο ευάλωτα κράτη-μέλη χρειάζονται στήριξη και πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των υποδομών. Χρειάζεται ε, ανάλυση των δυνατοτήτων που έχουμε, ανάλυση των περιφερειακών υποδομών, των υφιστάμενων υποδομών, προτού αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε νέες. Όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται ε, προσοχή στις υποδομές τους, ε, στην τιμολόγηση, ιδιαίτερα ε, για αέριο που φτάνει από τρίτες χώρες και επίσης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ε, σχέδια δράσης που έχουν προτείνει τα τρία, οι τρεις υψη, ομάδες υψηλού επίπεδου ε, ανά περιφέρεια, για τη Βαλτική δηλαδή, για την Νοτιοδυτική Ευρώπη και η ομάδα Κεντρικής Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Ε, πρέπει λοιπόν να τις ακούσουμε για την συνδεσιμότητα. Τώρα, αποθήκευση. Στόχος μου ήταν να ενισχυθεί η αποθήκευση και να δοθεί έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα ο κλάδος. Ε, δεν έχουμε την δυνατότητα να χάσουμε αυτούς, αυτούς ε, τους στρατηγικούς πόρους αυτή τη στιγμή. Διότι ήδη παρατηρείται ύφεση στα κέρδη της Βιομηχανία αυτή. Δεν μπορούμε τώρα να, να ανοικοκλίνουμε τους αγωγούς ανάλογα με το πότε θέλουμε περισσότερο ε, αέριο ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν στο σχέδιο έκθεση έχω προτείνει τρία μέτρα. Τα εξή. Καταρχά, αύξηση των προσπαθειών σε περιφερειακό επίπεδο για αύξηση τη αποθήκευση. ορισμενα ορισμένα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερε δυνατότητε αποθήκευση από κάποια άλλα και γι' αυτό θα πρέπει να ε, επιτευχθεί μια ισορροπία. Έπειτα, οι ε, κάτοχοι των ε, εγκαταστάσεων αποθήκευσης θα ε, πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε να υπάρχει είτε σωστή συντήρηση, είτε να υπάρχουν νέες, με, ε, νέα, νέες δυνατότητες αποθήκευσης στην αγορά. Έπειτα, η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για τους κώδικες μετάδοσης θα πρέπει να ε, ενισχυθεί με νέες προτάσεις για καλύτερη βελτιωμένη αποθήκευση. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήταν κάποια εισαγωγικά σχόλια. Όπως γνωρίζετε, αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο δηλαδή ακόμα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα για τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν να ε, τηρήσουμε όλο το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφε Γιώργη. Και τώρα θα δώσω το λόγο ε, στους σκιώδεις, πρώτο κύριο Τζανονάτο. Ευχαριστώ τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ανδρέας ε, Γιούρκο, με τον οποίο είχαμε την ευχαρίστηση να συνεργαστούμε. Τον ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας ε, που ξεκινήσαμε μαζί. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος, διότι ήδη έλαβε υπόψη τα γραπτά σχόλια τα οποία του είχαμε αποστείλει. Και πρέπει να πω, σε ορισμένα σημεία το κείμενο ήδη ε, ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις δικές μας προτεραιότητες. Αναφέρομαι κυρίως στην ανάγκη ε, να ε, υπάρχουν stranded assets, καθώς επίσης και διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στην απώλεια αποτελεσματικότητας Επίση, ε, Επίσης θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον, υπο, ε, ε, από τον συνάδελφο να αναφερθεί στον North Stream έτσι όπως τον είχαμε αναφέρει άλλωστε και σε προηγούμενο ψήφισμα του προηγούμενου Δεκεμβρίου στην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, επίσης, το θέμα του Network Code είναι ε, κάτι απαραίτητο. Επίσης, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία χρήζουν ε, ε, επιπλέον ε, επεξεργασίες, κυρίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όσον αφορά επίσης τους στόχους για, το, για τον άνθρακα, καθώς επίσης και για τους κλιματικούς στόχους για το 2030. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην διαφοροποίηση, αλλά και σε ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα το οποίο αρκούντος θα περιλαμβάνει τις ε, ε, εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ε, εγώ πιστεύω ότι πριν δημιουργήσουμε νέες υποδομές για την υγροποίηση του φυσικού αερίου θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να εκμεταλλευτούμε τις υφιστάμενες υποδομές και τις διαμεθοριακές δυνατότητες που κατά αυτή την έννοια παρέχονται. Με τον τρόπο από αυτό θα μπορέσουμε ε, ουσιαστικά να ανταποκριθούμε στην ε, ε, ζήτηση και την προσφορά. Επίσης θα πρέπει κατά την άποψή μου να προσθεθεί στον, στο κείμενο μία αναφορά στην ανάγκη ενεργειακής απόδοσης ε, σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ε, όσον αφορά τώρα την υποδομή ε, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ. Συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος υποστηρίζει τη θέση της Κομισιόν. Ωστόσο θα προτιμούσα το κείμενο να μην υπογραμμίζει απλώς τις δυσκολίες που αυτό ε, προκαλεί στην ε, ε, βιομηχανία αλλά να διαβρύνει περισσότερο το θέμα. Όσον αφορά τώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο ε, ε, είναι μια καλή εναλλακτική ε, λύση. Αλλά πιστεύω ότι καλό θα ήταν να πούμε ότι η στήριξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο δεν θα πρέπει να αποβεί προς ζημία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Φλάβιο, λέει η Πρόεδρος, ο συνάδελφος Στοτσενόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και θέλω να το τονίσω. Συμφωνώ απολύτως μαζί του, αλλά και η ομάδα μου, ECR. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ενεργειακή ε, αγορά και την ολοκλήρωσή της. Πολλά ε, από όσα προτείνει η ε, έκθεση μας βρίσκουν σύμφωνους και τα θεωρούμε πολύ λογικά για το ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τέτοιους θερματικούς σταθμούς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να έχουμε όλη πρόσβαση για να υποφελούνται όλες οι περιφέρειες και κάτι ακόμα πρέπει να τονιστεί. Ή δυνατόν η συνεργασία να είναι περιφερειακή, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε διαφοροποίηση των πηγών και απεξάρτηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, στο θέμα των τερματικών ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που λέει η έκθεση είναι ε, ότι θα πρέπει να έχουμε δυνατότητες αποθήκευσης για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις. Και εδώ ε, βρίσκω πολύ καλή τη γεωγραφική κατανομή των ταμιευτήρων. Χρειάζεται ισορροπία στην προσέγγιση μας Θέλω και πάλι να τονίσω πόσο καλή είναι η έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για τις ιδέες του, για τη συνεργασία του, για το πνεύμα προθυμίας που επιδεικνύει. Θα κάνουμε σίγουρα τροπολογίες για το γεωγραφικό ε, αυτό θέμα της κατανομής των ε, εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ο συνάδελφος, η συνάδελφος ε, Πουνσέτ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εμείς ε, από την ΑΛΤΕ έχουμε ε, αντιρρήσεις αναπόφευκτα όχι μόνο η έκθεση, αλλά γενικά ε, οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκινούν από ένα τελείω λάθος αξίωμα. Ποιο λάθος δεν γίνεται. Τι λένε τα αντικειμενικά στοιχεία στην Ευρώπη και μας δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου πάγια τα τελευταία έξι χρόνια 23% και πάνω. Και παρόλα αυτά εμείς εμένουμε στο φυσικό αέριο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μας έκθεση ε, με πείσμα λέει το ε, διαφορετικό, το αντίθετο. Και αυτό δεν είναι ένα και δύο χρόνια, είναι μια ιστορία δεκαετίας. Θέλω να σας δείξω αυτή τη γραφική παράσταση που είναι πάρα πολύ εύγλωτη. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτή τη μαύρη γραμμή που βλέπετε ε, εδώ είναι η πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά αυτές οι προβλέψεις που είναι προς τα πάνω ε, είναι διακεκομένες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αυτό που προβλέπει η Επιτροπή, λέει, ε, και έχει προβλέψει από το 2000, που έχουν πέσει τελείως έξω. Είναι τελείως ε, ανεδαφικά αυτά, ούτε κατά διάνοια δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Πού τα βρήκε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έκαναν λάθος ε, έτσι ένα-δυο χρόνια, δέκα χρόνια τώρα, τυχαία, υπέρ των πολιεθνικών. Τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει στο εσωτερικό της ε, στελέχη των πολυεθνικών που έχουν διεισδύσει, που έχουν παρισφρήσει και κάνουν ε, αυτές τις προβλέψεις δεν θέλω να πω ότι εσκεμένα γίνεται αυτό και συνειδητά, ας πούμε ότι κάνει λάθος. Ε, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι ε, παρατηρητές, αναλυτές από την αγορά να κάνουν τις προβλέψεις, γιατί οι υποδομές στη συνέχεια χτίζονται με δημόσια χρήματα. Αυτές οι υποδομές τι είναι, αυτές οι προβλέψεις που είναι και ε, εσκεμμένες, Έχουμε πάνω από 280 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα για το φυσικό αέριο, για μεροληπτικές προβλέψεις που αποκλείεται να ε, είναι αποδοτικές μέχρι να τις αποσβέσουμε μέχρι το 2025 τουλάχιστον. Για ποιο λόγο θέλουν να αυξήσουν πάνω από 58% τις εγκαταστάσεις ορισμένα κράτη-μέλη. Σήμερα έχουμε κάποιες υποδομές που δεν τις χρησιμοποιούμε, που δεν τις εξαντλούμε και μάλιστα μας ανισχύει πάρα πολύ ε, που αυτές οι επενδύσεις δεν απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς και μεσοπρόθεσμα τι θα κάνουν, θα φρενάρουν αποτελεσματικά τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που για μας είναι εκ των όνου Παράδειγμα, μια χώρα που είναι δικιά μου, που έχει επενδύσει η Ισπανία στην πρόσβαση ε, και, υπερβολικά στο φυσικό αέριο, με πάρα πολύ φουσκωμένα στοιχεία και προβλέψεις, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τέτοιο βαθμό στοιχηχών, τελείωσε το έργο, εγκαινιάστηκε και μετά έκλεισε κιόλας και άρχισε να κατεδαφίζεται. Εσείς πιστεύετε ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση φυσικού ε, αερίου και ποιος θα επενδύσει στις ανανεώσιμες, αν έχουμε κλειστές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, έχουμε 7 των αριθμών τερματικά, που υπο, ε, χρησιμοποιούνται μόνο στο 12% και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 25% ε, του δυναμικού. Τι τα κάνουμε όλα αυτά λοιπόν. Οπότε το πρώτο που πρέπει να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να της πούμε ότι η δουλειά της είναι να υπερασπίζεται τους καταναλωτές τους πολίτες και όχι πονηρά συμφέροντα ολιγοπολιακά. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας κάνει εντύπωση στην έκθεση είναι ότι δεν αναφέρει καθόλου, παρόλο που είναι πάρα πολύ πρόσφατο, ε, τελειώνει τελείω. Ναι, ναι, τελειώνω, αλλά είναι σημαντικά αυτά που έχω να πω. Ε, πουθενά δεν βλέπω την αηφορία και τη βιωσιμότητα. Πουθενά δεν βλέπω την κλιματική αλλαγή. Βιωσιμότητα μιλάει μόνο για το ορυκτό καύσιμο. Είναι δυνατόν το φυσικό αέριο και το βιώσιμο να είναι στην ίδια πρόταση. Αυτό είναι... Προσπαθούν να μας πούνε ότι το λιγότερο ε, ε, βρώμικο ορυκτό καύσιμο, λέει ο κύριος ε, ε δεν είναι βρώμικο, είναι από τα πιο βρώμικα. Δεν βγάζει διοξίδιο του άνθρακα, μεθάνιο παράγει, πουθενά δεν το λέτε. Ε, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται με το μεθάνιο, είναι το κόκκινο, εκπομπές μεθανίου. Ναι, πρέπει να τελειώνετε, λέει η πρόεδρος. Ε, με κίτρινο λοιπόν είναι το διοξίδιο του άνθρακα, εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα λίγο, αλλά 80 φορές πιο βλαβερό είναι το μεθάνιο. Η πρόεδρος διακόπτηκε, χτυπάει και το μικρόφωνο για να διακόψει την ομιλήτρια. Ε, Θέλουμε λοιπόν οι επενδύσει να περιοριστούν στι απολύτω απαραίτητε και να μην κάνουν μεγάλες business τα ολιγοπόλια και οι πολυεθνικέ. Ευχαριστώ πολύ. Να λούνται, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευσή του θα πρέπει οπωσδήποτε να αναχθεί ε, σε προτεραιότητα κλιματική και ενεργειακή σε σχέση ε, και με την ε, ασφάλεια του εφοδιασμού και την ενεργειακή απόδοση για τα επόμενα χρόνια και βεβαίως να ενταχθεί και στον ενεργειακό οδικό χάρτη. Η μείωση Ε, των ε, αερίων θερμοκηπίου κατά 90% οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, αναφερθεί και στην προκειμένη περίπτωση. Όπως το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναφέρει επανειλημμένα, υπάρχει μία σταθερά διογκωμένη εκτίμηση της ζήτησης του φυσικού αερίου. Ε, αλλά η ε, ζήτηση το 2013 ήταν κατά ε, κατά 23% λιγότερο, μικρότερη από το πικ που είχε φτάσει στο το 2000. Τα προγράμματα επενδύσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη και τους στόχους του 2010, του 2030. Εδώ διατρέχουμε τον κίνδυνο εγκαταστάσεων που θα υπολειτουργούν οι υποδομές για το υγροποιημένο φυσικό ε, αέριο. Ε, ε, είναι πολύ σε χρήση ενέργειας με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την χρήση τους η χρήση των, η εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2014 ε, ήταν μονάχα στο 13%. Ε, και θεωρούμε ότι ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε ε, με αυτές τις επενδύσεις τη στιγμή που τα, οι πόροι μειώνονται και η ζήτηση είναι ευθύνουσα. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο πολύ καλύτερο. Μπορούμε να αναπτύξουμε εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το φυσικό αέριο και εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιήσουμε τι ήδη υπάρχουσες δομές, καθώς επίσης και αρχές όπως η αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών και των ε, κρατών μελών το ε, αέριο παραμένει ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο ε, ε, δημιουργεί, το, το οποίο προκαλεί εκπομπές μεθανίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο επίσης σε πολλές περιοχές του κόσμου παράγεται μέσω της υδραυλικής ρογμάτωσης θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να ε, προχωρήσουμε σε ε, μία στοχευμένη μεταστροφή από τα ορυκτά καύσιμα και οπωσδήποτε να μειώσουμε τις επενδύσεις. Γι' αυτό, κύριο Ηλικιώτης. Εγώ αρχικά ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο τον Αντρασκού, για την δουλειά που έκανε, καθώς και για την προσπάθεια του να συμπεριλάβει στο πρώτο του κείμενο θέσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες. Η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αγροποιημένο φυσικό αέριο πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια μέσω τη καταπολέμηση τη ενεργειακή στόχια, τη διασφάλιση τη ισότιμη πρόσβαση στην ενέργεια για όλου, τη μείωση τη εξάρτηση από του αγωγού και τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού. Δεν μπορεί να παραβλέπουμε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περισσότερο περισσότερα από 100 BCM, κυρίω από τον Κατά. Ε, και είναι γι' αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σημαντικό να οι δερματικοί σταθμοί υγροποίηση να αξιοποιούν και τι εγχώριε πηγέ ενέργεια, ε, θέση η οποία ε, δυστυχώ απουσιάζει από την έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα του τι λένε κάποιοι συνάδελφοι, στι επόμενε δεκαετίε το LNG θα είναι το κύριο και το βασικό στην εμπορία του φυσικού αερίου διεθνώ και των θα περιοριστούν δηλαδή τα συμβατικά καύσιμα και αυτή είναι η πραγματικότητα που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο γιατί το LNG δημιουργά μια ευελιξία στην αγορά. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσθεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον αξιοποίηση των χώριων πηγών ενέργεια. Ε, έχω ω παράδειγμα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο στην Κυπριακή ε, ΑΟΣ και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει στην Κύπρο ένα κράτο μέλο, ε, τερματικό σταθμό υγροποίηση, η οποία θα αξιοποιά και τα κοιτάσματα τη ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, που είναι ε, ε κοιτάσματα πολύ σημαντικά για την ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια και τη τροφοδοσία ε, τη Ένωση και για να μπορούν έτσι να μειωθούν σημαντικά και οι περιφερειακές ανισότητες που υπάρχουν ε, κυρίως στα κράτη-μέλη της Μεσογείου. Ε, είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο για την επίτευξη του στόχου και τη άρση τη ενεργειακή απομόνωση, στην οποία βρίσκονται ε, καταδικασμένα κράτη και περιοχέ τη Ένωση. Ε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη στήριξη σε ευάλωτα κράτη για τη δημιουργία υποδομών. Να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν σήμερα κράτη όπω η Κύπρο, η Μάρτα, η Ιρλανδία, που χρησιμοποιούν 100% συμβατικά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ε, και ακριβώς πρέπει ε, σε αυτές τις περιοχές να προωθούν έργα κοινού ενδιαφέροντος ε, που είναι σημαντικά με αυτές τις απαραίτητες υποδομές να μπορέσουν αυτά τα κράτη να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές, τις, τον εφοδιασμό και να αρθεί η απομόνωση. Είναι γι' αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντική η αξιοποίηση μιας στρατηγικής για το LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ωραία. Πήραν το λόγο λοιπόν ε, οι σκιώδες Τώρα ο κύριο Κέλλη έχει εγγραφεί για να μιλήσει. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως ο εισηγητής μας έκανε μια πολύ καλή σύνοψη του πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι πρέπει ε, να γνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει το φυσικό αέριο. Αν πρέπει να έχουμε διαφορετικές πηγές ενέργειας, πρέπει να δούμε τις ε, ευκαιρίες που έχουμε και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μία από αυτές. Στην Ιρλανδία, τη δική μου χώρα, πολλές φορές λέμε ότι είμαστε ένα νησί γεμάτο ενέργεια. Τώρα έχουμε ε, φυσικό αέριο σε 20 χρόνια μέσω του νέου αγωγού που από το Ηνωμένο Βασίλειο θα είμαστε ανεξάρτητοι. Ωστόσο, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πού είμαστε, ξεκρέμαστε είμαστε όσον αφορά, όσον αφορά τον ε, ενεργειακό εφοδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν το ο τερματικός σταθμός ε, είναι κάτι που σχεδιάζουμε εδώ και χρόνια, αλλά μόνο χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιηθεί. Χρειάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αναγνωρίσει αυτήν την στρατηγική. Χρειάζεται μια ευρύτερη στρατηγική η οποία είναι προς το συμφέρον μας και πρέπει και εμείς να αναγνωρίσουμε τα ωφέλη της. Άκουσα αρκετούς που είπαν ότι η προσφορά και η ζήτηση του φυσικού αερίου μειώνεται. Στη δική μου χώρα όμως ε, η προσφορά μειώνεται για πολύ φυσικό λόγο. Δεν υπάρχει. πολύ ε, κρυώνουν, δεν υπάρχει θέρμανση, χρησιμοποιούμε άνθρακα και άκουσα εδώ να λένε ότι ο άνθρακας είναι πιο καθαρός από το φυσικό αέριο. Όμως, ε, εν ελήψη ανανεώσιμων πηγών, το φυσικό αέριο νομίζω είναι η προτιμότερη λύση και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της λύσης. Εάν ε, λοιπόν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε αυτούς τους τερματικούς σταθμούς, τότε δεν θα κάνουμε μόνο πολλά για τον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά και για την ενεργειακή ανεξαρτησία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μόζερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι επικεφαλής του τμήματος προμήθειας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε να μιλήσουμε και σε αυτό το σημείο. Καλωσορίζουμε την έκθεση του κυρίου ε, Γκιουρκ γιατί πιστεύουμε ότι έχει αδράξει τα κύρια στοιχεία και ενισχύει κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτά θα πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια της, ε, ε, των ε, μέτρων για, το, για την κλιματική αλλαγή 2030-2050. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε τους διεθνείς εταίρους μας έτσι ώστε να μην υπάρχει ή να μειωθεί η έκκληση μεθανίου. Εάν ε, οι όροι και οι προφυλάξεις λαμβάνονται σωστά, ε, τότε το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι πιο αποδεκτό από οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο στα πλαίσια, ε, όσον αφορά τη χρήση του, δηλαδή στα πλαίσια μιας ε, οικονομίας ε, με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Όσον αφορά τώρα τις εισαγωγές, η τάση είναι είτε, σταθερο, είτε σταθερή είτε ελαφρώς αυξητική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις σχετικές υποδομές. Πρέπει η εσωτερική αγορά να λειτουργεί σωστά έτσι ώστε το αέριο ε, το οποίο εισάγεται να προωθείται ε, απρόσκοπτα έτσι ώστε να συμβάλλει σε μια ε, οικονομία με λιγότερο άνθρακα. Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την χρήση των υπαρχουσών υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου καθώς επίσης και τις δυνατότητες αποθήκευσης χρησιμοποιώντας και υποδομές σε γειτονικές ενδεχομένω χώρες θα πρέπει να είναι επίσης απρόσκοπτη η μεταφορά η διασυνοριακή έτσι ώστε το σύστημα να είναι καλό ε, και ε, να αποβεί υπέρ εν τέλει των καταναλωτών ε, διότι το φυσικό αέριο οπωσδήποτε είναι λιγότερο βρώμικο από τον άνθρακα υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ε, καλό στοιχείο όσον αφορά την διαφοροποίηση και την ευελιξία. Παρέχει την δυνατότητα γρήγορης ε, ανταπόκρισης σε νέες ε, απαιτήσεις. Δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις σε σταθερές δομές και υφίστανται με τον τρόπο αυτό, υφίσταται με τον τρόπο αυτό λιγότερο ε, τις ε, ε, επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης γεωπολιτικής αστάθειας. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κλείσουν αποθηκευτικοί χώροι χωρίς λόγο ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μειούμενη ζήτηση για ε, αποθήκευση, αλλά θεωρούμε ότι η προσέγγιση της Κομισιόν είναι πολύ λογική και δεν χρειάζεται να ληφθούν βιαστικές αποφάσεις. Σε διεθνές επίπεδο πρέπει να εργαστούμε ε, στην οδό της συνεργασίας με άλλες χώρες έτσι ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα αλλά και να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ότι θα ε, υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης παροχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που με καλέσατε. Ευχαριστούμε ε, τον εισηγητή για την έκθεση και όλους για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μόζερ. Ο εισηγητής μας ε, θέλει σύντομα να κάνει κάποια τελικά σχόλια. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Και θα τα πάρω όλα στα σοβαρά. Ε, ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ένα από τα σχόλια που έκανα στην αρχή. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο και η αποθήκευση αυτού. Ε, σίγουρα Δεδομένε της ενεργειακές ανάγκες υπάρχει ο πειρασμό να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για την Ενεργειακή Ένωση. Πιστεύω όμω ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Ταυτόχρονα θέλω να σας διασφαλίσω ότι και εγώ θέλω να αποφύγω αυτήν την ενεργειακή εξάρτηση. Τώρα, να πω ότι έχω επίγνωση του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, μια στρατηγική για την αποθήκευση φυσικού αερίου και αυτή είναι πιο σημαντική για κάποια κράτη-μέλη από ό,τι για κάποια, κάποια άλλα. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν απόλυτη κάλυψη, κάποια μηδενική. Και είναι σαφές ότι οι χώρε οι οποίε έχουν μικρό ποσοστό διαφοροποίησης, Ιρλανδία, χώρες Βαλτική, Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, χρειάζεται ε, να δώσουμε έμφαση στην αποθήκευση του ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όμω, παρά τι διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη, είμαι πεπισμένο ότι όλοι μα θα υποφεληθούμε από την ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά ενέργεια, διότι η συνδεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω, και είναι προ το συμφέρον όλων μα. Και αυτό ε, συνεπάγεται και τη δημιουργία αποθήκευση για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τώρα, η επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουλίου, Δευτέρα, στο Στρασβούργο. Το, θα λάβετε τις συμβαστικές τροπολογίες εγκαίρως, αλλά αυτό εξαρτάται και από το πόσες τροπολογίες θα υποβληθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα τα πούμε με τους ε, σκιώδες στο Στρασβούργο και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω πολύ ε, κυρία Πρόεδρε σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο λίγη στις 12 το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και μετά, και μετά έχουμε τις άλλες προθεσμίες 11 Ιουλίου ε, για τη συζήτηση επί των τροπολογιών και Σεπτέμβριο η ψηφοφορία. Ολοκληρώσαμε να σας πω ότι στις 27 Ιουνίου της, στις Βρυξέλλες το απόγευμα και στις 4 ε, Ιουλίου το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία στην οποία ε, υπενθύμησε ο εισηγητής. Τελειώσαμε λίγο πιο πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ταχύτητα με την οποία πήρατε το λόγο. μπορούμε λοιπόν εδώ να αποχαιρετιστούμε και να πάμε να κάνουμε άλλα